στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Έχουμε εδώ πέρα ένα σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών και κύριε Μαρινέσκου έχετε ευθύ αμέσω το λόγο. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχατε τη δυνατότητα να μελετήσετε την, το σχέδιο εκδομοδότησης. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις. Εν γέννη θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν. Οι ε, πολιτικές ομάδες μου έχουν πει ότι θα υποστηρίξουν αυτές τις ε, συμβαστικές λύσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, πολιτικές ομάδες ε, το έχουν κάνει αυτό. Λοιπόν, τι ζητάμε. Ζητάμε μια αύξηση του προπολογισμού για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υποστηρίζουμε το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, το ΣΕΦ. Ζητάμε όμως ο μηχανισμός αυτός να επικαιροποιηθεί. Δεν θέλουμε νέο κανονισμό. Προκειμένου να έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον απαραίτητο χρόνο για να κλείσουμε το νομοθετικό αυτό σχέδιο μέχρι τις επόμενες ε, ευρω... Ε, ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον το ποσό που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια, γιατί ξέρετε ότι μειώθηκε εν συνεχεία κατά 27% Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μπορείτε να διαβάσετε στο σχέδιο γνωμοδότηση. Να σα πω πάντω ότι προτείνουμε να διευρύνουμε το ΣΕΦ και στι οδικέ μεταφορέ, διότι ξέρετε ότι είδαμε ότι θα ήταν θετικό να έχουμε έναν συντονισμό από την DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν οι 10 διάδρομοι και ο κεντρικός οδικός διάδρομος. Περισσότερο συντονισμό επίσης χρειαζόμαστε ή να έχουμε τουλάχιστον κάποιο συντονισμό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, από την DigiMove για όλα τα κονδύλια, διότι χρειαζόμαστε και εμείς καλύτερο συντονισμό, όπως γίνεται και με τα περιφερειακά ταμεία, για να μπορούμε και στον τομέα των μεταφορών να ολοκληρώσουμε τους διαδρόμους μεταφορών. Χρειάζεται επίσης συνέργεια και συντονισμός με τους εθνικούς προπολογισμούς, προκειμένου να κινούμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση και έπειτα έχουμε και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι συνέργειες μεταξύ των χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτά είχα να σας πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Ο κύριος Έρκτουκ τώρα και ο δισηγητής έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Morning. Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Ε, εξ ονόματος του κύριου Καπούτο, μια και δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα, να πω το εξή. Δεν έχω και πάρα πολλέ παρατηρήσει από πλευρά μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρνέσκου, που συμπεριέλαβε πιο πολλά από τα, στοιχεία, πιο πολλά από τα στοιχεία μα σε ό,τι αφορά την ε, συνδεσιμότητα. Και η πρόταση γενικά είναι αποδεκτή. Σα ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ ο κύριος Τσίλερ. Ευχαριστώ, Κάριμα. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Μαρινέσκου για την έκθεση αυτή. Ε, μερικά στοιχεία επιγραμματικά, γιατί το ECR υποστηρίζει τους πιο πολλούς συμβασμούς. Το ΣΕΦΕ θα πρέπει να συνεχίσει την χρηματοδοτητά και να αυξηθεί η χρηματοδότησή του. Τα χρηματοοικονομικά ε, μέσα όπω το ΕΦΣΙ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τι επιδοτήσει. Αυτά είναι σημαντικά για διαφορετικού λόγου, γιατί υπάρχουν κάποιοι τρόποι μεταφορών που είναι πιο ελκυστικοί για το ΕΦΣΙ και χρηματοδότηση μέσω του ΕΦΣΙ και υπάρχουν κάποιε διαφορέ ε, μεταξύ ε, χωρών και περιφερειών. Και φυσικά υπάρχουν και οικονομική και κοινωνική διάσταση στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την συνδεσιμότητα. Και σε ό,τι αφορά τα μέσα από την πολιτική συνοχή, θα πρέπει να αυξηθούν τα μέσα για την περίοδο μετά το 2020. Θα πρέπει να μειωθούν οι διαφορές και τα χάσματα στην συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών και οι οικονομικές διαφορές. Αυτό ήδη αναφέρθηκε υποστηρίζουμε, αλλά δεν θα υποστηρίξουμε τις ε, τροπολογίες για την μείωση του θορύβου, ούτε ασφαλώς την ειδική γραμμή για τον τουρισμό που θεωρούμε ότι αποτελεί πρόβλημα με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τελίντσικα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μαρινέσκου Με χαρά μου τον ευχαριστώ. Εν συντομία, τώρα με ενοχλεί ο κύριος Μαρινέσκου, εγώ τον ευχαρίστησα και αυτός να με ενοχλεί. Δεν με αφήνει να μιλήσω, πρόεδρε, πιο σοβαρά τώρα. Νομίζω ότι είναι καλή, καλές οι συμβαστικές τροπολογίες και εκτιμώ αφενός τη στρατηγική προοπτική προς το μέλλον και νομίζω ότι εκφράζουμε όλα όσα πρέπει να εκφράσουμε για τις μεταφορές μετά το 2020. Πέρα από την τρέχουσα θετία του Κοινοβουλίου, νομίζω ότι είναι καλή, καλό το ισοζύγιο μεταξύ όλων των στοιχείων. Κοιτάμε όλες τις πλευρές επαρκώς. Αναφέρθηκαν τα πιο επιτυχή οικονομικά μέσα, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και γενικότερα. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν προσδοκίες για αύξηση αυτών. Θεωρώ ότι αποτελεί γενικά αυτό μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ε, προσφάτως στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά υπάρχει σωστή κατάρτιση και κατάσταση πολιτικής. Ε. Και έτσι χωρίς δισταγμό θα προτείνω στην ομάδα μας να υποστηρίξει όλες τις συμβαστικές προτάσεις. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπας Έκχαουτ, θα ήθελα να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους του κυρίου Νίλσεν, μια ομάδα προσκεκλημένων από το Πανεπιστήμιο του Κέτεμπορκ. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Είσαστε νέοι και δυναμικοί. Ελπίζω λοιπόν σήμερα να ανακαλύψετε και διαφορετικά στοιχεία τα οποία θα σας χρησιμεύσουν στο μέλλον σας. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Έικαουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε νεαρή προσκεκλημένη από το Κέντεμπορ και ζητώ συγγνώμη που δεν είναι πολύ έντονη και ζωηρή η πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχουμε πολλά θέματα, αλλά και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Μαρινέσκου τον εσύ, γιατί προφανώς τώρα κοκκινίζει και είναι πολύ νευρικός που όλοι τον ευχαριστούν. Νομίζω ότι είναι καλή, καλές οι συμβαστικές προτάσεις, ε, όλες οι, όλα τα αιτήματα και οι απαιτήσει που ετέθησαν και από πράσινη πλευρά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τη χρηματοδότηση, το περιβάλλον, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί. Και νομίζω ότι από κοινού το κείμενο και η άποψη της Επιτροπής Μεταφορών είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά το επόμενο που Και θα υποστηρίξουμε λοιπόν ως πράσινοι τους εμειβασμούς για την υποδομή, για τις υποδομές Euroville. Φαντάζομαι ότι θα το υποστηρίξει η Επιτροπή παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και έχετε ακόμα όλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούγκριν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να... Θα ήθελα να υπάρχει ένας προϋπολογισμός όπου θα γίνονται τομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν καλά γιατί εξακολουθούν να προβλέπονται τόσο μεγάλες δαπάνες. Θα ήθελα πραγματικά να έχουν γίνει περικοπές ε, και σε ό,τι αφορά τις απώλειες ε, τις οποίες θα έχουμε όταν δεν θα συμπεριλαμβάνεται πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Van la parole est à vous. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Μπορεί να είναι λίγο βαρετό βέβαια που συμφωνούμε όλοι, αλλά έχω ένα σχόλιο. Ε, όπως ο κύριος Λούγκρεν, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Διαβάζοντας το συμβασμό 5, ε, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με την δήλωση αυτή ότι πρέπει να αυξηθεί το κομμάτι του προπολογισμού που αφορά τις υποδομές και τις μεταφορές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα υπάρξει μείωση ίσως και 50% της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και μια πιο έξυπνη χρήση ε, των ε, κονδυλίων, ίσως μέσω ενός επαναπροσανατολισμού ε, οι μεταφορές εδώ παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρει ο συμβιβασμός αυτός, αλλά με αυτή την ερμηνεία μπορώ να δεχτώ τον συμβασμό 5, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ταυτόχρονα, έτσι. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις χρηματοδότησης ε, στα πλαίσια ε, των περιορισμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και όχι απλώς να, απλώς να ζητάμε περισσότερα, διότι πιθανότατα θα έχουμε λιγότερα θα πρέπει να, όμως να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα, να έχουμε μια πολιτική ε, που να βασίζεται στην απόδοση και στον τομέα της πολιτικής συνοχής γενικότερα και όχι απλώς να ζητάμε περισσότερα χρήματα. Διότι αυτό δεν είναι και τόσο ρεαλιστικό. Υπάρχουν τρόποι να πετύχουμε τον στόχο μας ε, και εγώ ως συντονιστής ε, της Επιτροπής Ρέτζη θα το εξετάσω το θέμα αυτό διότι έχει ξαναγίνει αυτή η συζήτηση η πολιτική συνοχής μπορεί να εξυπηρετήσει και στόχους ε, στον τομέα των μεταφορών. Όταν μιλάμε τώρα για τις υπηρεσίες και την επέκταση των οπεδοτήτων τους, ε, έχουμε το λαμπρό παράδειγμα ε, της ε, του κανονισμού της ΕΑΣΑ, θα πρέπει να σκεφτούμε τη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την ΕΑΣΑ. Δεν μπορούμε να τους ζητάμε να έχουν αυξημένα καθήκοντα χωρίς να τους δίνουμε τα μέσα για να τα διεκπαιρεώσουν. Ευχαριστώ τον κύριο Φαν Μίλτεμπεργκ. Η Ιζαμπέλα Ντεμόντε έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παίρνω και εγώ το λόγο για να αναφερθώ περισσότερο στον τουρισμό. Θεωρώ δεδομένο ότι η Επιτροπή μα πρέπει να υποστηρίζει και τον τουρισμό. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να υποστηρίξουμε και τον κλάδο αυτό, που είναι τρίτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ένας κλάδος ο οποίος θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, μόνο ότι έχουμε γνωρίσει μια σημαντικότητα οικονομική κρίση σε πάρα πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνεται σημαντική μηνύα και στον τουρισμό στην γνωμοδότηση αυτή, καθότι θα πρέπει να επενδύσουμε στις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες, αλλά και στη βιωσιμότητα του κλάδου αυτού. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε και την δυνατότητα να αναπτύξουμε περισσότερο τον τουρισμό και στις πιο περιφερειακές ζώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι αναγκαστικά μόνο στις περιοχές της πόλης εκείνες που ήδη γνωρίζουν μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη που έχουν πιο κεντρική θέση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της οικονομικής ανάκαμψης στην οποία αναφερόμαστε στη γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να καλύπτεται και ο κλάδος τουρισμού καθότι μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκραπίνη έχει το λόγο. Δεν θέλει μάλλον το λόγο. Απλά την καρτούλα σας θέλατε, μάλιστα. Ε, θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να μας πει την απόψή της. Ο Λιβιέ Σιλά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή και όλες τις τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνες που υπογραμμίζουν την σημασία των στόχων της πολιτικής μεταφορών, ιδιαίτερα την ανάγκη να ολοκληρωθεί το ε, δίκτυο διευρωπαϊκών ε, μεταφορών, ε, την βελτίωση των ε, υποδομών και την απανθρακοποίηση των τομέα των μεταφορών και την ψηφιοποίηση επίσης. Βεβαίως ε, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι τα συγκεκριμένα ποσά στον προπολογισμό. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως σίγουρα καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Μαρινέσκου για να κλείσουμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τα καλά λόγια σε ό,τι αφορά την αύξηση του προπολογισμού τώρα. Ε, είναι σαφές ότι πρέπει να ζητήσουμε αύξηση του προπολογισμού. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να προτείνουμε και κάποια μέτρα τα οποία θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική την όλη προσπάθεια. Και αυτό είναι σαφές. Γιατί αυτή η πρόταση να ζητήσουν περισσότερα χρήματα από την ε, συνοχή. Είναι όντως μια θαραλέα πρόταση αυτή. Εγώ υποστηρίζω την πολιτική συνοχή, αλλά αυτή τη στιγμή ε, στην πολιτική συνοχή υπάρχουν πολλά project που αφορούν τις υποδομές μεγάλα project, ε, αυτοκινητόδρομοι, ε, σιδηρόδρομοι. Γιατί λοιπόν να μην τα βάλουμε αυτά στο ίδιο κεφάλαιο, ε, να συντονιστούμε για να συμπληρώσουμε και αυτούς τους διαδρόμους. Γιατί το καλύτερο για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι να συμπληρωθούν οι διάδρομοι των υποδομών. Ιδάλλως θα έχουμε ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εκεί. Δεν, υπάρχει, δηλαδή, δεν θα υπάρχει δηλαδή ένας πλήρης ολοκληρωμένος διάδρομος. Γι' αυτό Τώρα, με τον προπολογισμό θα γίνει μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να καλύψουμε το κενό του Brexit, ε, το κενό των νέων πολιτικών, άμυνα, ασφάλεια, μετανάστευση. Είναι αλήθεια αυτό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι ενδεχομένως κάποια κράτη-μέλη θα προτείνουν να είναι ίδιος ο προπολογισμός τουλάχιστον με το φετινό. Να ίδια τα ποσά. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε να φτάσουμε ένα, στο κατάλληλο επίπεδο προπολογισμού και να μπορούμε να προστατευτούν όλες τις πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο από τις 9. Πάμε στο επόμενο σημείο. Επιτάχυνση της καινοτομίας για καθαρή ενέργεια. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε και η συγκήτρια είναι η Ισαμπέλα Δε Μόντε. Η Ισαμπέλα Δε Μόντε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες. Να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους τους κοιόδης συγητές οι οποίοι έδειξαν πολύ επικοδομητικό πνεύμα και θεωρώ ότι καταλήξαμε σε πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις που ε, αντικατοπτρίζουν τελικά όλες τις διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν και όλα τα μέσα και τους τρόπους μεταφοράς. Έχουμε οκτώ συμβαστικές τροπολογίες συνολικά. Είχαμε και κάποιες συμβαστικές προτάσεις λίγο πιο τεχνικής φύσης, ιδίως όσον αφορά την τυπολογία ανανεώσιμων μορφών πηγών μάλλον ενέργειας. Παρ' όλα αυτά είχαμε και αρκετές τροπολογίες, ιδίως όσον αφορά το υδρογόνο και την ηλεκτροκίνηση, καθώς επίσης και τη διάρκεια της, ε, των συσσωρευτών και το πόσο θα μπορούσαμε, για, πιο μεγάλο, για πόσο πιο χρονικό διάστημα συγχωρείτε, θα μπορούσαμε να αποθηκεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, ηλεκτροκίνηση για τα λεωφορεία. Αναφορές επίσης σε νεοφυείς ε, επιχειρήσεις γίνονται στροπολογίες, καθώς επίσης και δυνατότητα επένδυσης σε νέες ε, μορφές οικολογικές ενέργειας. Πάρα πολλέ τροπολογίε αναφέρονται σε κάποιε δυσκολίε που έχουμε ακόμα στον τομέα των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ακόμα μια σημαντική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο των μεταφορών και ο τομέας των μεταφορών παραμένει ένας από τους βασικούς λόγους ρήπανσης των πόλεων. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη Συμφωνία των Παρισίων για τις κλιματικές αλλαγές. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να δίνουμε νέες κατευθυντήρες γραμμές για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, για τις δυνατότητες αποθήκευσης και για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνουμε όλο και πιο συγκεκριμένε αναφορές στην γνωμοδότηση αυτή όσον αφορά τις καθαρές μορφές ενέργειας και αναφερόμαστε στην ολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, τη χρησιμοποίηση του υδρογόνου και το καθεξής. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τους συναδέλφους οι οποίοι υποστήριξαν τις συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. αντικαθιστώ τον συνάδελφο τον κύριο Κλούνε που ταξιδεύει από την Ιρλανδία προς την υπηρετική Ευρώπη είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό το θέμα της υπήρου και το πώς συνδέεται με τα νησιά ε, θα ήθελα λοιπόν καταρχήν ε, να μεταφέρω τα συγχαρητήρια της κυρίας Κλούνε προς την κυρία Τελμόντε όπως και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης αλλαγής. Πρέπει οι μεταφορές να γίνουν πιο καθαρές. Η ενέργεια γενικότερα πρέπει να γίνει πιο καθαρή. Εγώ όταν ήμουν στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο ε, θεωρούσα ότι η ανάγκη αυτή είναι και απειλή για, τον, για τη βιομηχανία αλλά έμαθα εδώ στην Ευρώπη ότι είναι και ευκαιρία. Ε, μην αποσταθεροποιείτε τον κύριο Βαντενκάμπ. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Στην ομοδότηση της κυρίας Δελμόντε, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των αναγκών του κλάδου και την ανάγκη καινοτομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε βεβαίω περαιτέρω, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη γενικότερη ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Η τρίτη συνιστόσα εδώ είναι η ψηφιοποίηση. Χρειαζόμαστε καινοτομία και εδώ στην καινοτομία μπαίνει το θέμα της ψηφιακής εποχής. Η γνωμοδότηση πάντως είναι πολύ ισχυρή, πολύ καλή και εκ μέρους της κυρίας Κλούνε θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη ψηφοφορία αύριο στην κυρία Ντελμόντε. Εμείς θα υποστηρίξουμε πάντως ε, τους συμβιβασμούς, τις συμβαστικές απολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, του έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις τροπολογίες. Λέει ο το Σενόσκι δεν είναι εύκολο η επαγγελματική χρήση των μεταφορών μέσω της καινοτομίας ε, είναι ένα ευρύ ζήτημα. Αφορά πολλά και διάφορα, ε, πολλές και διάφορες πτυχές, ε, πολλές από τις οποίες είναι τεχνικές. Ο τομέας των μεταφορών έχει τεράστιες δυνατότητες ε, βελτίωσης ε, σε ό,τι αφορά την αποδοτική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών. Δεν πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι το να πετύχουμε τους στόχους στον τομέα της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας είναι κάτι το οποίο θα περιπλέξει τα πράγματα σε επίπεδο περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ε, ενδεχομένω ε, να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων παγκοσμίω. διότι τα πράγματα εκεί δεν είναι απλά. Τώρα, ο συσχετισμός μεταξύ των, της έρευνας, ε, της καινοτομίας και της ψηφιαποίησης στον τομέα των μεταφορών είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται Βεβαίω οι επενδύσει σε τομέα αυτό χρειάζονται σταθερότητα, χρειάζονται μακροπρόθεσμη, ε, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, διότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε ένα πεδίο ανοιχτό σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό ε, στα προγράμματα, προγράμματα έρευνα ε, μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε οι λίγοι πόροι που έχουμε να μην σπαταλώνται. Ε, πόροι πολύ σημαντικοί για την έρευνα και την καινοτομία. Εμείς θεωρούμε οι αλλαγές στον τομέα των μεταφορών μας πάνε προς τεχνολογίες ε, με μικρότερη χρήση ενέργειας, μικρότερη χρήση ενέργειας προσανατολισμένες προς τους ε, καταναλωτές, με πολύ πιο γενικευμένη ψηφιοποίηση με βάση τους στόχους που μας, έχουν, μας έχετε παρουσιάσει εδώ, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα την τεχνολογική ουδετερότητα, διότι δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ποια κατεύθυνση ακριβώς θα πάρει η πρόοδος. Αναμένουμε νέες τεχνολογίες σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας, τις μπαταρίες, ε, είναι σαφές ότι η παρούσα τεχνολογία δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ε, αναμένω με τη μονησία της συζητήσης με την εισηγήτρια. Με βέβαιος ότι θα συζητήσουμε σε, ένα πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο όχι ο κ. Στερλίτσκα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου του, συναδέλφου του ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Στο όνομά του λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ντελμόντε, Ντεμόντε ε, για την καλή και ισορροπημένη αυτή την γνωμοδότηση. Επίσης ο συνάδελφος εκτιμά ιδιαίτερα το, τη συνεργασία ε, που της προσέφερε και ως συγγητές ή ε, συγγήτρια. Ε, σύμφωνα με τον συνάδελφο η γνωμοδότηση αυτή αποτυπώνει ε, πιστά το αίτημά μας να μειωθεί, να μειωθούν οι ε, ανισότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή, μεταξύ των αστικών κέντρων και της υπαίθρου και μεταξύ βεβαίως των πιο αναπτυγμένων περιοχών και εκείνων που είναι πιο πίσω σε επίπεδο υποδομών και ποιότητας υποδομών. Εμείς υποστηρίζουμε τους στόχους της Κομισιόν να δοθεί προτεραιότητα και να προωθηθούν project ε, αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και να δοθούν σχετικά κίνητρα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στον τομέα των μεταφορών αυτό περιλαμβάνει βεβαίω και τον τουρισμό. Έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη συζήτηση αυτό. Να επικεντρωθούμε προς ε, ε, projects για καθαρό, καθαρή ατμόσφαιρα όπως ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η χρήση ηλιακή ενέργεια, υπάρχει βεβαίω και το θέμα τη τεχνολογική ουδετερότητα με το οποίο συμφωνούμε. Τέλος να πω ότι η Άλντε θα υποστηρίξει όλες τις προτάσεις συμβασμού, τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι ισορροπημένο, επαναλαμβάνω, το κείμενο και εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι όλες οι τροπολογίες που υποβάλαμε απο, αποτυπώνονται, εκπροσωπούνται στην τελική γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Monsieur la parole est à vous. Ε, Ο κ. Σανταλούντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Τιμόντα και τους υπόλοιπους και ε, για την πολύ καλή συνεργασία και οι συμβαστικές προτάσεις περιλαμβάνουν τα πιο σημαντικά στοιχεία και όλες τις ε, συμβαστικές προτάσεις, ε, όλες τις τροπολογίες που είχαμε προτείνει, γι' αυτό λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να κοστίζουν παραπάνω και οι εκπομπές θα πρέπει λοιπόν τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιηθούν και για την πράσινη μετάβαση. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να προωθούν τις καινοτομικές αυτές αλλαγές. Και αυτά όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και να την ανακόψουμε, αλλά θα μας καταστήσουν και πιο ανταγωνιστικούς, προκειμένου να είμαστε οι νικητές από τη νέα αυτή τεχνολογία και από την πράσινη αυτή μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τελούντε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Λούγκριν θέλει να πάρει και αυτό το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Ντεμούντα για την γνωμοδότηση και νομίζω ότι αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειάζεται αλλαγή. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν από κάποια χρόνια ήδη. Είχαμε για παράδειγμα αντιμετωπίσει το θέμα των εκπομπών των φορτηγών. Αν συγκρίνουμε τι γινόταν πριν από 15 χρόνια σε ό,τι αφορά τις εκπομπές των φορτηγών, τα πράγματα προφανώ έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ στην Σουηδία. Ε, υπάρχει, αν θέλετε, ε, μια δοκιμαστική απόσταση στους αυτοκινητοδρόμους που χρησιμοποιείται ηλεκτρικό μόνο. Είναι σημαντικό λοιπόν να, κοιτάξουμε και θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Εδώ υπάρχει τεράστιο δυναμικό. για τη μεταφορά επίσης και των ε, προϊόντων, για τις ροές των ε, προϊόντων. Δεν είναι ακόμα εντελώς αποτελεσματική και αποδοτική η μέθοδος μεταφορών αυτών. Υπάρχουν λοιπόν ε, ελλείψεις ό,τι αφορά το συντονισμό. Αν υπήρχε μεγαλύτερος συντονισμός και γεμίζονταν καλύτερα τα φορτηγά, θα γλιτώναμε και πάρα πολλές εκπομπέ σα. Ευχαριστώ και πρόκειται πραγματικά για ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κραπίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να συζητήσουμε αυτή την πολύ σημαντική ε, γνωμοδότηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισαμπέλ, αλλά και τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε προφανώς την καινοτομία, την οικολογική, τις οικολογικές ε, μεταφορές. Θα πρέπει να βρούμε λύσει ε, για να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και να βρούμε και οικονομικά μέσα. Γιατί προφανώς ε, χρειάζονται χρήματα και επενδύσει. Χρειάζεται ενερμόνιση λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι οι τοπικέ αρχέ έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, καθώ οι αστικέ μεταφορέ και για παράδειγμα οι δημόσιε συγκοινωνίε αποτελούν μεγάλο τμήμα, μεγάλο, μεγάλη πηγή εκπομπών και λοιπόν Θα πρέπει νομίζω κυρίως να υπογραμμίσουμε τις οικολογικές μεταφορές. Ένα παράδειγμα αν σε όλες τις πόλεις μας ε, θα μπορούσαμε να καταδείξουμε πόσο υποστηρίζουμε τις καθαρές μορφές ενέργειας. Σκοπός μας είναι να υπάρχει πραγματικά καθαρή ενέργεια στον τομέα των μεταφορών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γραπίνη και τώρα να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσω το λόγο στον κύριο Ζόμπι. Thank you, Madam Chair. Κύριε. Λοιπόν, ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή τη γνωμοδότηση. σα ακούμε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει την Επιτροπή σας για τις προτάσεις της. Χαιρετίζουμε τη γνωμοδότηση αυτή, γιατί θεωρούμε ότι οι προτάσεις που κάνει συνάδουν απόλυτα με τα όσα προτείνουμε και εμείς στην δική μας σχετική ανακοίνωση, καθώς επίσης και στο θεματολόγιο έρευνας και κοινοτομία για τις μεταφορές. Τα όσα προτείνεται στη γνωμοδότηση αυτή ενισχύουν τελικά τις δικές μας προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταφέρουμε μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών να εξυγχρονίσουμε τις μεταφορές και να καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε τον απότερο στόχο μας που είναι ανταγωνιστικές καθαρές μεταφορές χωρίς αποκλεισμούς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Ντεμόντ, έχετε το λόγο προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα μέσω της γνωμοδότησης αυτής, μια γνωμοδότηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα για τα σημεία αυτά τα οποία προωθούμε προς την άλλη Επιτροπή. Ιδίω όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους. Δεν ήταν εύκολο να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές απόψεις των πολιτικών ομάδων. Παρόλα αυτά σήμερα είδαμε ότι στην πράξη είναι δυνατό κάτι τέτοιο και όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πλέον έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κλάδο το βιομηχανικό και τους υποστηρικτές του περιβάλλοντος και της ενεργειακής βιωσιμότητας, γι αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της βιομηχανίας είδαμε όλο και περισσότερες ευκαιρίες στον τομέα της καινοτομίας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τους συναδέλφους και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε αύριο να υπερψηφίσουμε την γνωμοδότηση αυτή, αλλά μου φαίνεται ότι ήδη αυτό θα συμβεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεμόντε. Αύριο θα ψηφίσουμε στις 9 η ώρα το πρωί. Θα διακόψω τώρα τις εργασίες μας προκειμένου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση που όλοι περιμένουμε. σε σχέση με το Brexit και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον τομέα των χερσαίων μεταφορών. Να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας. Στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας για τη δημόσια ακρόαση. Λοιπόν, Κάνουμε διάλειμμα 15 λεπτών. Στις 10 πάντως θα ήθελα να είστε στην αίθουσα για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ακρόαση, παρακαλώ. Η Επιτροπή μας σήμερα οργανώνει μία ακρόαση δημόσια για τις επιπτώσεις του Brexit ε, στις χερσαίες μεταφορές. Ο στόχος αυτής της ακρόασης είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, υψηλού επίπεδου ε, του τομέα των σιδηροδρόμων και των οδικών μεταφορών για να καταλάβουμε καλύτερα να προλάβουμε οι δυνατόν τους ενδεχόμενους κινδύνους ε, που εμφανίζονται με την αποχώρηση του Μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε Επίσης πως οι εταιρείε αυτών των δύο μεγάλων κλάδων ε, προετοιμάζονται για την αλλαγή αυτή και ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, ε, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη δουλειά τους, δίτρα ό,τι αφορά τις μεταφορές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Επίσης θέλουμε να γνωρίζουμε τι αναμένουν από τις, από ε, ε, οι εκπρόσωποι του κλάδου. Σε δύο σκέλη θα, θα χωριστεί η συζήτηση. Πρώτα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, τριών ενώσεων ε, οδικών μεταφορών και το δεύτερο κομμάτι θα αφορά μια συζήτηση με τους εκπροσώπους ε, των σιδηροδρόμων. Λοιπόν, το κάθε πάνελ θα συνοδεύεται από ερωτήσεις, από συζήτηση με τα μέλη μας. Ε, βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να καλωσορίσω το σύνολο των ομιλητών και τώρα θα ήθελα να κάνετε μια μικρή παρουσίαση για το θέμα. Ξεκινάω το πρώτο πάνελ που αφορά τις οδικές μεταφορές και με μεγάλη χαρά έχω δίπλα μου εδώ την Βερόνα Μέρφη που είναι η πρόεδρος ε, του Irish Roads, Road Haulage Association. Μαζί μας είναι επίσης ε, ο κύριος Χούκαμ, ο οποίος είναι ε, επικεφαλής του Freight Transport Association, καθώς και τον Daniel Kern από την IRU. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις οδικές μεταφορές. Λοιπόν, είναι αρκετά απλά τα πράγματα σε ό,τι τη διαδικασία. Ο καθένας έχει 7 λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους ε, βουλευτές. Και μετά βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Ξεκινάμε με την κυρία Μέρφη. Για 7 λεπτά. Καλή σας μέρα. Το όνομά μου είναι Βερόνα Μέρφυ. Άρχισα να οδηγάω 19 ετών φορτηγό και 20 ετών άνοιξα την εταιρεία μου μεταφέροντας τον εαυτό μου από την Ιρλανδία στην Ιταλία. Αυτό πριν, πριν πάνω από 25 χρόνια, έξω ότι έχουν αλλάξει πολλά. Εξακολουθώ να μεταφέρω κρέας από την Ιρλανδία στην Ιταλία για τους ίδιους πελάτες. Ε, τέσσερα 4 με 6 φορτηγά είναι ε, το αριθμό για μικρέ εταιρείε, για τι μεγάλε όμω φτάνει, και, φτάνει τι εκατοντάδε. Εγώ του εκπροσωπώ όλου. Ε, Όπω τα γνωρίζετε, μόλι ε, περάσαμε από τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία τη χώρα μα και κατευθείαν περνάμε στο Brexit. Η Ιρλανδία είναι η μόνη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χερσαία σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, τα χερσαία σύνορα με την Βόρεια Ιρλανδία ε, Σημαίνει ότι η Ιρλανδία θα είναι ένα νησί εντό ενό νησιού όταν, Ευρω... όταν το νοσίλιο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τραγικέ επιπτώσει ενό σκληρού Brexit για την Ιρλανδική οικονομία και δίδρα για τον συγκεκριμένο κλάδο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ε, είναι, έχει, Μιλάμε για 5.000 θέσει εργασία, 2,5% ε, της απασχόλησης ε, στην ελληνική οικονομία. Τα περισσότερα μέλη μας ε, ζουν στην Ήπεθρο και οι θέσεις εργασίας αυτές είναι πολύτιμες. Ο κλάδος αυτός επίσης προσπαθεί να στείλει σημαντικά αγαθά σε επιχειρήσεις και στους ανθρώπους ένα μεγάλο ποσοστό των φορτηγών μεταφέρει προϊόντα τοπικά επίσης ε, είναι πραγματικά ο αιμοδότης ε, της εμπορικής ζωής. 1,2 ε, εκατομμύρια αξίας προϊόντων μεταφέρονται από, το, από την Ιρλανδία στο Μένο Βασίλειο. Οι επιπτώσεις του Brexit είναι ήδη απτές, διότι άμεσα έχουμε μία απειλή για την βιωσιμότητα λόγω της ε, αστάθειας ε, που συνδέεται με τον Brexit, έχει αποδυναμωθεί η λίρα, υπάρχει νευρικότητα στην αγορά. Αν είναι σκληρό το Brexit, το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχουν σύνορα μεταξύ ε, της υπηρετικής Ευρώπης ε, και του Ινωμένου Βασιλείου και μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Θα είναι πιο υψηλά, υψηλή και οι δασμοί και αυτό θα αυξήσει το κόστος. Τα φορτηγά που θα περνάνε τα σύνορα ενδεχομένως να τους ζητείτε να... Ε, να ακολουθούν μια διαδικασία που ακολουθούνταν πριν την ενιαία αγορά. Ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν επίση ε, δασμοί η τέτοιου είδου ε, περιορισμοί θα οδηγήσει σε καθυστερήσει στι μεταφορέ αυτέ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν οι επιχειρήσει να μεταφέρουν, να μετακινήσουν το κόστο αυτό στου καταναλωτέ, διότι θα αυξηθεί η τιμή, θα μειωθούν οι καταναλωτέ μα. ήδη τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα, και θα βρεθούν πολύ εκτός ε, δουλειάς. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια υποδομή που να επιτρέπει γρήγορη και αποτελεσματική μετακίνηση, ε, ασφαλή στάθμευση. Η τεχνολογία πρέπει να μας βοηθήσει για να έχουμε μια πλήρη ψηφιο, πλήρως ψηφιοποιημένη τελωνιακή διαδικασία. Για να προγραμματιστούμε όμως σωστά είναι πολύ σημαντικό ο τομέας των μεταφορών και οι απόψεις τους ε, υπόψη του να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ο τομέας αυτός να ενημερώνεται έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίσουν το μέλλον τους και όχι απλώς ε, να περιμένουν πότε θα πέσουν από τον κρεμό. Ε, πολύ λίγα ξέρουμε ακόμα για τη φύση αυτού του Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα, η Ιρλανδία πρέπει να προστατευθεί και όποια μέτρα παρθούν ενδιάμεσα που θα επηρεάσουν την Ιρλανδία θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα προσεκτικά. Παραδείγματο χάρη η εισαγωγή του πακέτου για την κινητικότητα θα αλλάξει θεμελιωδώς το πώς εργάζονται οι οδικοί μεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά έχουν θεσπιστεί με βάση το status quo, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη το Brexit. Πώς λοιπόν να τόσο ε, πλήρες πακέτο μπορεί να προχωρήσει χωρί να γνωρίζουμε επακριβώ ε, ποιε θα είναι οι επιπτώσεις της αποχώρησης τη Ηνωμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να την προσέχει και να την βοηθάει ώστε ε, να μπορέσει να μειωθεί, να μπορέσει να μετριαστεί η ανταραχή και να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου. Ε, το πακέτο αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή θα, θα δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα, θα δημιουργήσει μια πραγματική καταιγίδα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ε, αλλά και οι εργαζόμενοι επηρεάζονται πάρα πολύ από την οδηγία για, την, ε, για τον χρόνο εργασίας, τα διατάξεις που αφορούν κυρίως την υπηρετική Ευρώπη και τις ανάγκες της ήδη είναι μη ευελεκτροσύστημα δεν ταιριάζει σε χώρες όπως η Ιρλανδία, ε, διότι να μην ακολουθούμε τη θαλάσσια οδό για να φτάσουμε στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο ο τομέα των οδικών μεταφορών είναι στην πρώτη γραμμή τη της οικονομική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδία και στην πρώτη γραμμή ε, τη σχέση μεταξύ Ιρλανδία και Υπηρετική Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκοί θύνοντε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η ζωτική σημασία συνιστόσα τη Ιρλανδική και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζωή θα προστατευτεί στο μέτρο του δυνατού. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει μια δέσμευση ότι ο κλάδος μας ε, θα διέπεται από ασφάλεια, από ένα ασφαλές περιβάλλον ε, και δεν πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει περαιτέρω κόστος ε, τουλάχιστον για 36 μήνες έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν την δύσκολη εποχή για την Ιρλανδία και τις επιχειρήσεις μας. Ως μεταφορέας εξετάζοντας το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του πακέτου κινητικότητας βλέπω ότι η επιπτώση για την Ιρλανδία ε, με βάση το Brexit δεν, έχουν ληφθεί, δεν έχει ληφθεί υπόψη. Είναι ένα πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ιρλανδία. Εγώ είμαι μια επιχειρηματία που εκπροσωπώ ε, του εργαζόμενου μου. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να σα ζητήσω να λάβετε υπόψη σα τι επιπτώσει ε, του Brexit, ιδιαίτερα να συζητάτε το πακέτο για την κινητικότητα. Δεν πρέπει να αφήσετε την Ιρλανδία πίσω, να μην την ξεχάσετε ω μια ξεχασμένη γη ε, στι ακτέ τη Βρετανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη αυτή παρέμβαση, παρέμβαση ιδιαίτερα στεναρή θα έλεγα, ιδιαίτερα σαφής, με ένα ηχηρό μήνυμα που ζητά από εμά, ευρωβουλευτές, να λάβουμε τις ευθύνες μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Κύριε Χούκμαν, εσείς έχετε τώρα το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα το πρωί. Ονομάζομαι James Hookman. Είμαι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, FTA. Είναι η μεγαλύτερη τέτοια ένωση με 17.000 μέλη που μεταφέρουν εμπορεύματα όχι μόνο μέσω των οδικών μεταφορών αλλά και μέσω των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, επίσης μεταφορών και νέων μεταφορών. Συμμετέχουμε σε διάφορους οργανισμούς, εκπροσωπούμαθαν επίσης και στο Δουβλίνο και έχουμε δημιουργήσει επίσης το Παγκόσμιο Φόρουμ Φορτωτών, Πρακτόρων και Μετακόμισης. Συμμετέχουμε επίσης στη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρακτόρων και Μετακόμισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι Βρετανοί εισαγωγοί και εξαγωγείς θεωρούν ότι ε, ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και επίσης μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ από το Brexit. Το Brexit θα δημιουργήσει νέα σύνορα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερους ελέγχους, σε νέες απαιτήσεις στα σύνορα και αυτό ενδεχομένω να παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η κλίμακα του εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε. Το μέγεθος εμπορίου λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί περίπου σε 8 φορές το μέγεθος του εμπορίου που έχουμε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Περίπου 185.000 επιχειρήσεις θα καλούνται πλέον να υποβάλουν τελειωνιακέ διασαφήσει, καθώς επίσης και άλλες διατυπώσεις στα σύνορα για πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, ένα 80% περίπου των οδικών μεταφορών που εκτελούν τη διαδρομή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 27 υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το ζήτημα του Brexit δεν αφορά σίγουρα μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τρεις βασικούς ε, Παράγοντες που θα επηρεάσουν τη μελλοντική εξέλιξη του εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ θα προκύψουν σύνορα μετά το Brexit και θα επηρεάσουν τι νέε απαιτήσει που θα έχουμε πλέον όσον αφορά το εμπόριο. Θα έχουμε όμω και σημαντικού κινδύνους όσον αφορά την διαθεσιμότητα ποσοστώσεων για τα οχήματα ή τις άδειες των οχημάτων να περνούν πλέον τα σύνορα και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το ζήτημα των προσόντων, την αναγνώριση των προσόντων μάλλον των οδηγών. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα επί την οποία θα θέλαμε να έχουμε διευκρινήσει όχι μόνο από την κυβέρνηση του Μένου αλλά και από τι κυβερνήσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε λοιπόν ότι μα απασχολεί πάρα πολύ η διασύνδεση και η βασική εμπορική δρόμη η εμπορική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μάνου Βασιλείου αλλά και του Μάνου και Ιρλανδίας. Πολύ φοβάμαι ότι με τα νέα σύνορα τα οποία θα προκύψουν, θα προκύψουν και πάρα πολλέ μεγάλε καθαστερήσει, πολύ μεγάλε ουρέ στα σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει πραγματικά καθόλου χώρο στα λιμάνια προκειμένου να συσσωρευτούν όλα αυτά τα οχήματα, όλα αυτά τα φορτηγά. Χώρος δεν υπάρχει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στον Βασίλειο, ούτε στην Ιρλανδία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να προκληθεί τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το λιμάνι του Ντόβερ εκτίμησε ότι κάθε επιπλέον δύο λεπτά καθυστέρησης με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν θα προκαλέσει ουρά 27 χιλιόμετρων και φαντάζεστε ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και στο Καλέ και κατά αναλογία και σε άλλους λιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιρλανδίας. Η πρόκληση λοιπόν είναι πολύ μεγάλη για το Μάνο Βασίλειο, αλλά εξίσου μεγάλη είναι και για τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω για τι κυβερνήσει τη Γαλλία, του Βελγίου, των κάτω χωρών, τη Ισπανία και βέβαια τη Ιρλανδία. Θα προκύψουν νέε τελωνιακέ διασαφίσει, οι οποίε θα πρέπει πλέον να συμπληρώνονται Ξέρουμε ότι έχουν αρχίσει ήδη ορισμένε χώρες να προσλαμβάνουν ε, νέο προσωπικό επιβολής του νόμου στα σύνορα και θα έχουμε επίσης 300 ε, εκατομμύρια επιπλέον διασαφείς που θα πρέπει να υποβάλλονται στα νέα σύνορα που θα προκύψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα προκύψουν πολλά νέα προβλήματα. Όσον αφορά την ε, ομαλή συνέχιση της, ε, του εμπορίου και της μετάβασης των οχημάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ζήτημα των ε, αδειών. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε πλέον ελεύθερη κυκλοφορία των φορτηγών και ενώ σε άλλους τομείς υπάρχει δυνατότητα αναδίπλωση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δεν προβλέπεται θέση αναδίπλωση όσον αφορά τι ε, εμπορευματικέ ε, οδικέ μεταφορέ. Έχουμε το σύστημα ECMT, το οποίο δεν μπορεί να ισχύσει όμω στο μέλλον, και αυτό γιατί οι ποσοστώσει προβλέπονται αντιστοιχούν μόνο στο 5% των, του υφιστάμενου όγκου πολίσεων. Βλέπετε ότι ο όγκος αυτός πολίσεων και ο αριθμός μεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου είναι τέτοιος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί το σύστημα ECMT της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών. Νομίζω λοιπόν ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσαρμοστούν πλέον στις αλλαγές που έρχονται για το μέλλον με το Brexit. Και τονίζω για άλλη μια φορά ότι ο κίνδυνος είναι κοινός και για τις δύο πλευρές και όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια ανάλογη κατάσταση υπάρχει και στις υδροδρομικές μεταφορές. Δεν θα καλύψω πάρα πολύ τον κλάδο αυτό, φαντάζομαι ότι στο επόμενο πάνω το καλύψετε περισσότερο. Είναι σημαντικό πάντως να συνειδητοποιήσετε ότι ανάλογες διευθετήσεις θα πρέπει να γίνουν και για τις συνδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, καθώς επίσης και για την αναγνώριση των προσόντων των οδηγών των τρένων. Θα ήθελα να συνοψίσω τα βασικά συμπεράσματα της ε, παρουσίασής μου αυτής λέγοντας ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα προκύψουν νέες ανάγκες για ελληνικέ διασαφήσεις και νέοι έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει να επιβληθούν, όχι μόνο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και οι υπόλοιπε κυβερνήσεις από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβουν δράση και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί επίσης και μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κλάδο των εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Προφανώς θα πρέπει οι μελλοντικές διαδικασίες που θα προκύψουν να αποτελέσουν αντικείμενο απλούστευσης. Θα πρέπει σε μια πρώτη φάση όμως να εγγυθούμε την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τονίζω για άλλη μια φορά ότι τα προβλήματα αυτά τα οποία προκύπτουν και που μα περιμένουν στο μέλλον αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο για τον Μανοβασίλειο αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σα που προφανώ ε, αναφέρει στοιχεία αριθμητικά τα οποία μα προκαλούν λίγο. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Με τον κύριο Κέρν. Έχετε το λόγο και εσείς για 7 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και που με προσκαλέσατε. Ντάνιελ Κέρν ονομάζομαι και εργάζομαι για την IRU, για την ε, οργάνωση ε, χερσαίων οδικών μεταφορών. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στην διαφάνεια υπάρχουν ε, χώρες με μπλε χρώμα με ενεργό συμμετοχή σήμερα και αρχικά πρόκειται για μια οργάνωση με αποτύπωμα Δυτικής Ευρώπης. Αυτό προκύπτει από τις χώρες που έχουν σημειωθεί με μοβ χρώμα στο χάρτη για την κινητικότητα στην Ευρώπη. Στοιχεία της Eurostat, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Γιατί, γιατί μας δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος. Όχι μόνο οι οδικές μεταφορές, αλλά γενικά οι μεταφορές και μιλάμε για ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αύξηση μέχρι το 2050 σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. η μεταφορά 60% στα εμπορεύματα, 40% και πλέον στους επιβάτες. Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη λοιπόν, ένα αναπτυσσόμενο κλάδο Πρόκειται για ένα κλάδο που μετράει στην Ευρώπη και θα επηρεαστεί από τον Brexit. Οι προτεραιότητε τη IRU στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρει. Όπω φαντάζεστε, το πακέτο κινητικότητα τη Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση είναι υψηλά στην ατζέντα μα. Brexit και μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη χρήση άνθρακο. Τι περιμένουμε λοιπόν και τι δεν θέλουμε, τι δεν επιθυμούμε να προκύψει από το Brexit ως IRU τώρα υπάρχουν έγγραφα τοποθετήσει τα οποία και δημοσιεύτηκαν σήμερα. Εστιαζόμαστε στην πρόσβαση στην αγορά και στα τελωνιακά ζητήματα και άλλα θέματα θα θέλαμε να επεξεργαστούμε και να ε, κοιτάξουμε, όπως για παράδειγμα κοινωνικές συνθήκες, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κάποια βασικά στοιχεία τώρα σε ό,τι αφορά το Brexit. Στο IRU έχουμε μια ομάδα εργασίας η οποία ηγείται, αν θέλετε, της διαδικασία σχηματισμού απόψή για το Brexit. Το να μην υπάρξει συμφωνία δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Σε καμία περίπτωση θα θέλαμε να διατηρηθεί τουλάχιστον το status quo στη μεταβατική περίοδο. Πού και πού μας προσογγίζουν διάφοροι και μας ε, ρωτάνε τι δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να συμβεί σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την προσβασία στην αγορά. Οποιοδήποτε σύστημα ποσοστώσεων θα αποτελούσε μεγάλη στρέβλωση τη αγορά Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την πρόσβασή τη στην αγορά από πλευρά ΗΠΑ Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον λοιπόν του Brexit δεν ξέρουμε ακόμα γιατί ω τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αποδεκτό το κεκτημένο, να μεταφερθούν όλα στην εθνική ομοθεσία. Είναι η πρώτη όμως χώρα που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε λοιπόν σίγουροι και ενδεχομένω να πρέπει να δείξουμε μια κάποια δημιουργικότητα, μια κάποια ευελεξία στο τελική ανάλυση για την εξέβρεση λύσεων. Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες σήμερα στην αγορά σε ό,τι αφορά τα τελωνιακά ζητήματα, τις τελωνιακές διθετήσεις. Για παράδειγμα, η περίπτωση της Τουρκίας, πρώτη εναλλακτική λύση την οποία εξετάσαμε. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια μερική τελωνιακή ένωση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι οικονομία και η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο των G20 και έχουν και χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόμοια τα πράγματα και για την Ορβηγία, παρά το γεγονός ότι εδώ είναι μεγάλη εναρμόνιση των τολυνιακών διαδικασιών και διεκπαιρεώσεων. ελέγχονται από τους Νορβηγούς ή τους Σουηδούς ε, συναδέλφους ε, τα φορτηγά και αυτή η δυνατότητα αποκλείστηκε λόγω της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το θέμα και η περίπτωση της Ελβετίας. Η ελβετική λοιπόν περίπτωση είναι ενδιαφέρουσα. είναι μέρος του FTA από το 1972. Τώρα σήμερα έχουμε περίπου 100 συμφωνίες που θα ρύθμιζαν σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολε οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία και η εφαρμογή και η υλοποίηση. Αυτό διατείνονται κάποιοι άλλοι πάλι στα κράτη-μέλη δηλώνουν ότι είναι μια πολύ ευέλικτη λύση αυτή που τελικά έχει εξευρεθεί. Το πλήρες διαζύγιο τώρα, αυτό θα είναι το πιο στρεβλωτικό, αν θέλετε, σενάριο μετά το Μάρτιο του 2019. Η, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έμενε ως ανεξάρτητη χώρα. Φυσικά θα δεσμεύονταν ακόμα από τις κανόνες και τις προδιαγραφές των διεθνών οργανώσεων, αλλά αυτό είναι το σενάριο το οποίο δεν προτιμούμε. Και να έχουμε υπόψη ότι είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό θα ενοχλούσε πάρα πολύ τη λειτουργία μας. Πρόσβαση στην αγορά. Δεν θέλουμε ποσοστώσεις, θέλουμε να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια με τη μερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία για τις οδικές μεταφορές γνωρίζοντας ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι και πιο ευρύε αυτέ αυτές οι διαπραγματεύσεις, αυτές οι συμφωνίες. Δεν θα χρειαζόταν έγκριση σε σχέση με ένα σύστημα ποσοστώσεων σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ε, αγαθών. Και εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση να μην υπάρξει συμφωνία σε ό,τι αφορά δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία περίπτωση θα χρειαζόντουσαν 27 ξεχωριστέ συμφωνίε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 27 κρατών μελών, κατά κερματισμό περιττό προφανώ. Και κλείνοντα, ποια είναι τα βασικά μα μηνύματα. Πέντε. Πέντε μηνύματα. Θέλουμε να είναι ομαλή η κίνηση οδικών μεταφορών μετά τον Brexit μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. σε μια επαρκή μεταβατική περίοδο όπου θα διατηρηθεί το status quo, πρόσβαση στην αγορά χωρίς ποσοστώσεις αλλά με ποιοτικά κριτήρια και πάλι και, μίας, και είμαστε μία, ένας κλάδος οικονομικός που βασίζεται βασικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να υπάρξει επιπλέον γραφειοκρατία μετά το Brexit. Και επίσης το νομικό πλαίσιο να είναι προβλέψιμο και ασφαλές. Να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Στο σημείο αυτό κλείνω την παρουσίασή μου και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και για τις τρεις παρεμβάσεις σας. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα απλά να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους της συναδέλφου της κυρίας Κλούν, που είναι εδώ μαζί μας. Καθώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, δεν ξέρω που κάθεστε βέβαια ακριβώς, μάλλον στο βάθος, πάντως καλώς ήρθατε. και μετά τις παρεμβάσεις σας αγαπητοί συνάδελφοι θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι παρεμβάσεις σας έτσι ε, μας πιέζουν κάπως. Είναι σαφή αυτά που λέγεται, αυτά που λέτε και, και επίσης είναι σαφές ότι επίγει ε, το ζήτημα αυτό. Αναφερθήκατε στο πακέτο για την κινητικότητα από το οποίο εργαζόμαστε. Ε, μας είπατε επίσης ότι πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο διοικητικό επίπεδο, διότι είναι πολύ βαρύ, με άμεσες επιπτώσεις ε, ε, στις μεταφορές. Ε, μας λέτε, ζητάτε μεταβατική περίοδο. Να πω βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις ε, εμείς προσπαθούμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και να λάβουμε υπόψη μας αυτό που μας λέτε. Λέτε κυρία Μέρφη το πακέτο κινητικότητας να, να ε, επιβραδυνθεί και να λάβει υπόψη ε, τις επιπτώσεις του Brexit. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό, διότι όντως είναι πολύ σημαντικά τα θέματα. Να ξεκινήσει όμως η συζήτηση Πρώτα ο κύριος Μάρκους Πίπερ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή αυτή εισαγωγή. Όντως, αντιμετωπίζετε και περιγράφετε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τεράστια. Ε, κοιτάξτε, ούτε εμείς ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και δεν είχαμε φανταστεί ότι θα καταλήξουμε και εδώ. Και τώρα με 20% των διοικητικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολούμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Brexit. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό αποτελεί ένα θέμα το οποίο το έχουμε συνδέσει με τεράστια ενόχληση. Ξετυλίγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την λύνουμε αντί να ασχολούμαστε με το μέλλον και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είμαστε πολύ ενθουσιώδεις. Σήμερα χθες ε, ακούσαμε ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να συνάψουμε εμπορική συμφωνία με την, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Ε, και οι δικέ σα παρεμβάσει προ την κατεύθυνση αυτή κινούνται. Θα ήθελα να θίξω δύο σημεία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Καταρχά, η μαγική λέξη ψηφιακά σύνορα. Ε, Τεχνολογίε blockchain, δεν θα μπορούσε όμως η τελική ανάλυση το σύνορο της ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου να αποτελέσει ένα προκάτοχο, αν θέλετε, μια τεχνολογική ευκαιρία η οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ε, σε άλλα μέρη για να τεθούν, αν θέλετε, όροι και ορόσημα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση οι μεταφορέ ρυθμίζονται κυρίω από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό δεν ικανοποιεί απαραίτητο πάντα όλου, γιατί πολλά πράγματα θεωρείται ότι είναι περιβολικά και θα σα επιβαρύνουν. Στο δικό σα το κλάδο υπάρχει αυτό το περίφημο cherry picking, δηλαδή την επιλογή α, αυτών που μας αρέσουν και το να αφήνουμε αυτό που δεν μας αρέσουν. Δηλαδή αυτή η ρύθμιση μας αρέσει. Τα ωράρια για παράδειγμα, οι ώρες ανάπαυσης, σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπλοκη νομοθεσία ή αποδέχεστε τη δική μας νομοθεσία α, ως έχει. Αυτό ασφαλώς ήταν και καλό επιχείρημα για την Μελλοντική Εμπορική Συμφωνία και για να καταλήξουμε σε μια προπαρασκευαστική λύση των συντομότερων δυνατών. Αν δηλαδή, αν εμείς ακούγαμε από εσά ότι κοιτάξτε εμείς ως ε, κλάδος μεταφορών ε, έχουμε επιβάρυνση, αλλά ως ε, μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης. Ε, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα, μας, θα ακολουθήσουμε αυτή την νομοθεσία. Άρα το θέμα των ψηφιακών συνόρων και το θέμα αυτό που σας ανέφερα σχετικά με την επιλογή ή όχι μεμονωμένων διατάξεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έτουκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από δική μου πλευρά. Η οχι μονομενων διαταξεων σας φράση, κυρία Μέρφη, Νομίζω ότι αποκρισταλώνει το δήλωμα ότι ως Δημοκρατία της Ιρλανδίας ε, δεν θέλετε να γίνετε ξεχασμένη χώρα. Ως σοσιαλιστές πρέπει να σας πω ότι φυσικά αυτό θα το αποτρέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί φυσικά είσαστε υπέρ της Ευρώπης. Και στέκει αυτό που είπε ο συνάδελφος Πίπερ, ότι τώρα τα πράγματα δεν εξαρτώνται από εμά. Ε, αν εξαρτάται από εμά, οι λύσει δεν θα είναι τόσο δύσκολε προφανώ. Το θέμα είναι ότι προφανώ ότι εμεί είμαστε εξαρτημένοι, γιατί ουσιαστικά αυτοί που κάνουν τι διαπραγματεύσει για τον Brexit είναι άλλοι. Μπορούμε προφανώ να απλοποιήσουμε κάποια πράγματα και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι θέλουν τι θέλει ο και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι, και το ακούσαμε αυτό, δεν είναι δυνατόν να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε από την νομοθεσία, από όλο το θέμα του Brexit και να προσπαθήσουμε να τα διαπραγματευτούμε για να αποδυναμώσουμε το σύνολο της συζήτησης, γιατί αυτό όντως αποτελεί λίγο cherry picking, όπως αναφέρθηκε. Δεν είναι όμως αυτό που επιθυμεί η Ευρώπη των 27. Και να θυμόμαστε ότι η απόφαση που θα κληθούμε να λάβουμε σε δύο χρόνια θα έχει φυσικά και επιδράσεις ενδεχομένω και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ομολογώ ότι είναι εντυπωσιακά τα αριθμητικά στοιχεία και προφανώς δεν θέλουμε επιπλέον γραφειοκρατία. Εννοείται ότι δεν επιθυμούμε ε, επιπρόσθετες ε, τελωνιακές και να προκληθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στους δρόμους. Αλλά παρόλα αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου θα πρέπει να γεννηθεί και θα πρέπει να δηλώσει τι είναι διατεθειμένη να κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει να παίρνει μεμονωμένες νομοθεσίες και να ξεκινάει ε, ξεχωριστή διαπραγμάτευση και αυτή η, αυτό το αίτημα για μεταβατική περίοδο. Αυτή η μεταβατική περίοδο κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει. Αλλά δεν θα βοηθήσει η μεταβατική περίοδος αν δεν έχει βρεθεί μια γενικότερη λύση για το σύνολο των ζητημάτων. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή ακρόαση είναι σημαντική για μα για να ξέρουμε τι δεν επιθυμείτε. Ποσοστώσει, μα είπατε, επιπρόσθετε ηλεκτρονικές ε, προδιαγραφέ, ε, γραφειοκρατία, και το ότι θέλετε προβλεψιμότητα και νομική ασφάλεια. Είναι προφανές. Αυτό θα το πολεμήσουμε. Αλλά, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι στη δική μας πλευρά. Η εθνική κυβέρνηση δεν μας ε, διευκολύνει. Σας ευχαριστώ, δική Πρόεδρε. Η κυρία Φώστρα έχει το λόγο. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές πληροφορίες που μας έδωσαν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που ελέγχθηκαν ε, από την κυρία Μέρφυ ε, όχι μόνο για το πακέτο κινητικότητας το οποίο είναι πολύ σωστό που το ανέφερε διότι είναι εξαιρετικά πλήρες πακέτο ε, και σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ το Brexit υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς όπου υπάρχουν διάφορα προβλήματα όταν προέρχεσαι από ένα νησί. Στην Επιτροπή Απασχόλησης, η οδηγία ε, για τις ώρες εργασίας, και τις ώρες οδήγησης, ε, είναι και άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν, διότι όταν κάποιος μεταφέρει αγαθά μέσω θαλάσσια οδού, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που είπε ο κ. Χούκαμ και τα σχόλιά του, Νομίζω ότι μας δώσετε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, ε, στοιχεία για το κόστος και αναφερθήκατε στις δεξιότητες των ε, ε οδηγών που βρισκόμαστε στη συνορικό επίπεδο σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από τη Βρετανική κυβέρνηση τουλάχιστον ότι σκοπεύουν να αλλάξουν τους κοινωνικούς κανόνες προς το χειρότερο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια. Ε, Επίσης ζητήματα όπως ε, τα προσόντα των οδηγών ή άλλα σχετικά ζητήματα δεν νομίζω να αλλάξει. Δεν είναι απαραίτητο, Ξέρω αν κάποιος το κάνει επίτηδες. Ε, και εμένα. Έχουμε πολύ καλά πρότυπα στον Εμένο Βασίλειο και εγώ ως πολιτικός ε, θα φροντίσω ε, να μην υπονομευθούν και δεν έχω τέτοιες ενδείξεις από, το, από την κυβέρνηση τουλάχιστον. Ε, επίσης σε επίπεδο Ενωμένου Βασιλείου υπάρχει ένα lobbying με τους υπουργούς μεταφορών ε, στα Υπουργεία του Ενωμένου Βασίλειο και εδώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο τρίτος ομιλητής ο κ. Κέρνης πρέπει να βρούμε λύσεις γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις ε, εξετάζουμε το κόστος ε, για το εμπόριο, για την απασχόληση βεβαίως όλα αυτά ισχύουν ε, εγώ τώρα δεν θέλω ούτε σκληρά σύνορα ε, με δασμούς. Δεν είναι αυτή η θέση μας, ε, κάτι το οποίο το ξέρετε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει όλοι μαζί ε, να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει κάθε, κάθε χώρα να προσπαθήσει να έχει μια ειδική μεταχείριση. Πρέπει στο τέλος της διαδικασίας και οι 27 αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο να οδηγηθούν σε, μια δίκαιη, σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα και τα πράγματα να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο ομαλά. Είναι σαφής ο στόχος αυτός και μπορούμε να τον πετύχουμε Επίσης ε, θα πρέπει οι ενώσεις, οι εμπορικές, τα επιμελητήρια, οι βιομηχανικές και αυτές να προτείνουν λύσεις. Οπότε συνεχίστε να κάνετε να, να, να ασκείτε πιέσει, να κάνετε lobbying. Εγώ, πόσο ξέρω, είστε πολύ αποτελεσματικοί. Συνεργάζομαι με πολλού συναδέλφου ε, ε, στα Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι είστε πολύ ενεργοί. Είναι πραγματικά εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση σήμερα και από Ιρλανδική πλευρά χαίρομαι που είστε εδώ, διότι εδώ μπορούν και οι πρόσωποι των άλλων 27 να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστεί αυτή η ελεύθερη ροή αγαθών, ε, εμπορίου, απασχόλησης. Μπορεί να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ την κυρία Φώστερ. Ο κύριος Τελίτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστούμε και για αυτές τις εξαιρετικά διαφορετικές παρουσιάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να επαναλάβω ε, αυτό που ελέγχθη ήδη σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Αυτή η Επιτροπή είναι σαφής. Ε, εμείς ακούμε και σκεφτόμαστε υπάρχουν και πολλοί ε, αυτό που θα, πρέπει, που να είναι εδώ βέβαια είναι οι Βρετανοί Υπουργοί Βρετανοί βουλευτές ε, και σε αυτούς που να απευθυνθείτε. Σε ό,τι φορά την Ιρλανδία τώρα βεβαίως αναγνωρίζουμε απολύτως αυτό το πρόβλημα και σας υποστηρίζουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το σχόλιο που κάνατε όμως για το πακέτο κινητικό, για την κινητικότητα. Ακούστε, δεν είμαι βέβαιος ότι συμμερίζομαι την άποψη της Προέδρου ότι μπορούμε να το καστερίσουμε. Ακούστε, αυτή τη στιγμή είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Το πακέτο περιλαμβάνει ε, μια σειρά από μέτρα εθνικά και δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει. Ε, υπάρχει κάθε συμφέρον να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα με το πακέτο και την κινητικότητα, έτσι ώστε να έχουμε νομική ασφάλεια, να έχουμε συνέπεια, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο έδαφος και όχι επιμέρους ε, σε κάθε κράτος μέλος. το θέμα είναι ποια τα στοιχεία του πακέτου τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις σε εσά. Αυτά ενδεχομένως να τα εξετάσουμε, να δούμε πώς αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη, να αντιμετωπιστεί με τροπολογίες, τροποποιήσεις, μια μεταβατική περίοδο ενδεχομένως, ε, διευκολύνσεις, ε, κάποια επιμέρους στοιχεία. Ε, θα ήταν καλό να ξέρουμε ποια είναι αυτά βέβαια από την πλευρά σας. Σε ό,τι αφορά και πάλι τις επιπτώσεις για μένα είναι σαφή τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι σαφέ. Ό,τι και να συμβεί τώρα έω την πραγματική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, αναγκαστικά θα χρειαστεί μια μεταβατική περίοδο. Ε, αν μιλήσουμε τώρα για τρία χρόνια, ε, πραγματικά αμφιβάλλω αν και αυτό είναι διαχειρίσιμο. Ακόμα και αν αρχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις σύντομα, είναι, ξέρετε, κάτι που παίρνει χρόνο. Έτσι λοιπόν, ε, όπως είπε η κυρία Φώστερ, ε, πρέπει να υπάρξει lobbying ε, είναι κρίσιμο, διότι δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, δεν αντιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας που θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο γίνεται πιο καλό ή να μειώσει τέλο πάντων του κραδασμού. σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του λόμπινγκ, καλό είναι να ξέρουμε και ποια, ποια είναι η ανταπόκριση. Ε, ξέρω ότι είναι πολιτικά δύσκολο να πει κανείς ότι θα αποτελέσουμε μέρος της ενίας αγοράς, αλλά πώς βλέπετε, ε, ποιες είναι οι, οι αντιδράσεις ε, σε ό,τι αφορά το λόμπινγκ που κάνετε για την Τελωνιακή Ένωση, παραδείγματος χάρη, ε, και ένα ερώτημα για την Ιρλανδία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Το πολιτικό είναι τα ανοιχτά σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας για μια σειρά λόγους. Ε, υπάρχει συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής, ε, θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα, έτσι. Και από τη δική σας ε, προοπτική, κυρία Μέρφη, εσείς πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να έχουμε σχόλ, ε, η σύνορα Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας ή Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Αναφέρομαι τώρα για το εμπόριο μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα για την υπηρετική Ευρώπη υπάρχει και η θαλάσσια οδός. Ευχαριστώ κύριε Τελίτσκα. Ε, ήθελα απλώς να διορθώσω κάτι, αν δεν με καταλάβατε καλά, για το πακέτο για την κινητικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούν να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα. Το πακέτο για την κινητικότητα έχει ξεκινήσει. Θα σεβαστούμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, στα πλαίσια του πακέτου κινητικότητας, όπως είπατε κι εσείς, ε, να κάτσουμε να σκεφτούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για σας, αυτό βεβαίως θα συμβεί. Αλλά για το χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. Να προσπαθήσουμε λίγο να το μαζέψουμε όμως. Ε, διότι καλό είναι να ακούσουμε και τις απαντήσεις από το πάνελ. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, συμμετέχοντες στο πάνελ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις που κάνανε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δικές σας αναδυόμενες προτεραιότητες. Θα ήθελα λοιπόν στον καθένα από εσά να θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο οποίο έχετε καταλήξει. σε περίπτωση που εγκαταλείψει το Μένο Βασίλειο και την Τελωνιακή Ένωση, κάτι το οποίο θα συμβεί ίσως τον Απρίλιο του 2019, τι σχέδια εσείς καταρτίζετε αυτή τη στιγμή εκ των προτέρων για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή. Ποιες διευθετήσεις προβλέπετε ότι θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν, ιδίως σε σχέση με τα Ιρλανδικά σύνορα γιατί εγώ φαντάζομαι θα προκύψουν μια τεράστια σειρά προβλημάτων και δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές της μάχης που να γνωρίζουν τελικά ποιες είναι επιπτώσεις και ποιο είναι τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέλιορ Λουνγκριν. Να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ πέρα την ε, κυρία Μάρφη, την οποία την ε, γνωρίζω από το παρελθόν. Εγώ πριν από 30 χρόνια ασχολούμαι ακριβώς με τον τομέα αυτό των εμπορευματικών μεταφορών και είμαι θα έλεγα ο πρώτος οδηγός φορτηγού που εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρίσκομαι εδώ από το 2014 και μετά. Εργάστηκα πολύ λοιπόν στα πλαίσια των οδικών διεθνών εμπορευματικών μεταφορών Ακούσαμε διάφορες εναλλακτικέ και υποθέσεις. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα δεν έχει παγιώσει μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit. Από παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει ακόμα να δει πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και βέβαια δεν έχουμε καν συνέλθει από το σοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σοκ τη απόφαση ε, του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε πώ θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση και ιδίω για τον τομέα των μεταφορών πώ θα λειτουργήσουν στο μέλλον τα πράγματα. Ξέρετε ότι ε, κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαμε όντω σύνορα και δασμού μεταξύ των κρατών μελών. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα τελωνία τα οποία θα προκύψουν τώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Θα θυμάστε ότι στο παρελθόν όταν δεν υπήρχε τελωνιακή ένωση και όταν υπήρχαν όντω τελωνιακοί έλεγχοι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις στα σύνορα. Πρέπει να καταφέρουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα αυτά στο μέλλον. Ευελπιστώ ότι ε, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε τελικά σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι θα ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις και ότι θα καταλήξουμε τελικά σε διευθετήσεις οι οποίες θα είναι θετικές, αν μη τι άλλο, για το δικό μας τον τομέα, το τομέα των μεταφορών. Και μην ξεχνάμε επίση ότι το μέσα αυτό έχει μια πολύ έντονη πλέον διεθνή διάσταση. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Η στρατηγική λοιπόν που θα ακολουθήσουμε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις διεθνείς μεταφορές. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε καταλήξει σε κάποιες εναλλακτικέ, αν έχετε μια συγκεκριμένη προτίμηση υπέρ της μίας ή της άλλης και πώς θα καταφέρουμε τελικά όντως να επιλύσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα το οποίο διαφαίνεται στο μέλλον. Υπάρχει plan B, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πρόεδρος, Όντως πραγματικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν όντω έχετε προετοιμαστεί για αυτό το οποίο προμηνύεται στο μέλλον. Μας δώσατε αριθμητικά δεδομένα τα οποία ακούγονται τρομακτικά, ιδίως ε, όσον αφορά τον όγκο και το μέγεθος των πωλήσεων, αλλά και όσον αφορά όλες αυτές τις νέες διατυπώσεις και διασαφείς που θα προκύψουν ε, μέσω των ε, νέων τελειωνιακών συνόρων που θα προκύψουν. Όπως είπε και ο κύριος Λαγκρίν, εσείς μεταξύ σας έχετε έναν κάποιο προκαταρκτικό οδικό χάρτη σε περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας για τον Brexit. Ο κύριος Πίπερ εν συνεχεία αναφέρθηκε σε αυτά τα ψηφιακά σύνορα. Πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Ο κύριος Σέρτουκα αναφέρθηκε στο ζήτημα της ε, απώλειας του κέρδους ε, που ενδεχομένως να πλήξει την δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αναφερθήκατε επίσης στο πακέτο κινητικότητας ε, και το αν θα μπορούμε τελικά να έχουμε μια μεταβατική περίοδος προς αυτό, αλλά πάλι δεν το αποφασίζουμε εμείς αυτό. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με αξιωματούχους, με αρμοδίους της Βρετανικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, για να, για θίξετε το, το ζήτημα αυτό της μεταβατικής περίοδου. Και ακούσαμε και ένα ακόμα ερώτημα, πολύ σημαντικό και αυτό, για την ε, κατάσταση που θα προκύψει για τους ίδιους τους οδηγούς, για τους επαγγελματίες του τομέα. Τι θα γίνει από επαγγελματικής, κοινωνικής πλευράς, αν ε, βγούμε από το νομικό αυτό πλαίσιο το οποίο εφίσταται αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά από το ενωσιακό δίκαιο. Δίνω δύο λεπτά στον καθένα για να απαντήσετε σε ερωτήσεις αυτές και μπορούμε να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και να προχωρήσουμε σε επικοδομητική ενταλλαγή απόψεων. Η κυρία Μέρφη έχει πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μας θέσατε. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για το πακέτο κινητικότητας, κατανοώ. Αλλά δεν νομίζω ότι από πρακτικής πλευράς οποιοδήποτε μου έχει θέσει το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Φυσικά και μπορούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι αντιμετωπίζουμε τεράστιο όγκο οδηγών και ο κανονισμό υπό τον οποίο λειτουργούμε είναι επαρκή. παρά το γεγονός ότι υπάρχει φυσικά συζήτηση για το κοινωνικό dumping και το πώς ε, περνάνε και αναπαύονται στα φορτηγά του οι οδηγοί. Κοιτάξτε, δεν του έχουμε δεμένους. Ε, στο τιμόνι τους ανθρώπους αυτούς. Κάνουν ό,τι θέλουν ε, με το χρόνο τους. Ε, και εγώ χτες ε, πήγα σε ένα ξενοδοχείο, 300 ευρώ πληρώσα, υπερβολικό, και ήμουν σε ένα ξένο δωμάτιο, σε ένα ξένο χώρο, με κακό μαξιλάρι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό, δηλαδή, για τον οδηγό να οδηγεί μετά από δύο νύχτες που έχει ξενυχτήσει. Αυτό είναι το πρακτικό θέμα. Το άλλο θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το ξενοδοχείο και τελικά θα το επομιστεί ο οδηγός. Όλα αυτά είναι πτυχές του πακέτου κινητικότητας. Κανείς όμως δεν κοιτάει τελικά τι ισχύει, ποιες είναι οι πρακτικές λύσεις. Κανείς ε, δεν ρωτάει τους οδηγούς. Ο τρέχον κανονισμός ε, για τους ταχογράφους είναι πραγματικά πάρα πολύ μειονεκτικός για μια χώρα νησί όπως ε, η Ιρλανδία. Θα μας πάρει μια μέρα παραπάνω να πάμε να έρθουμε στην υπηρετική Ευρώπη λόγω του Brexit. Αυτό είναι καλό. Κακό για μας ε, και κακό για όλη την Ευρώπη, γιατί τελικά χάνει ο καταναλωτής, χάνει το προϊόν, την αξία του. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρξουν αυξήσει ε, στις πωλήσει. Θα πούμε πάλι σε ύφεση. Αν κάποιος με ρωτούσε λοιπόν ποιο είναι το σχέδιο επαναχώρησης, θα ήταν να γίνω ευρωβουλευτής, να την πουλήσω την εταιρεία και να γίνω ευρωβουλευτής. Αυτό είναι το καλύτερο, γιατί δεν ε, βλέπω, κύριε Τέιλερ, τι ακριβώ θέλετε να κάνω ω μεταφορέα, τι να κάνω με τις διαδικασίε αυτές, γιατί συνεχίζονται ακόμα τα λόγια. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι το πακέτο κινητικότητας θα προκαλέσει ακόμα πιο πολύ μεγάλη ζημιά μετά τον Brexit και η Ιρλανδία θα είναι η χώρα που θα πληχθεί χειρότερα από το, την βορειοδυτική πλευρά της Ιρλανδίας για να φτάσουμε στην Υπηρετική Ευρώπη έχουμε να περάσουμε τέσσερα σύνορα. Πώς τα συγκρίνουμε λοιπόν αυτά με την Ελβετία. Αυτοί ένα σύνορο περνάνε. Τέσσερις φορές λοιπόν πρέπει να περάσουμε σύνορα. Κάτι τέτοιο πραγματικά είναι επώδυνο για τα άτομα τα οποία α, και στα τελωνία δεν θα είναι και σωστά εκπαιδευμένα, γιατί κανείς δεν έχει τέτοια εκπαίδευση για να λάβει τελωνιακά καθήκοντα. Όλοι οι κανονισμοί όπως οι ταχογράφοι ήδη καταρτίστηκαν το 2006, όταν δεν υπήρχαν σύνορα. Τώρα θέλετε οι ίδιοι οι κανόνες να ισχύουν με σύνορα, αλλά τελικά αυτός που επηρεάζεται είναι οι Ιρλανδοί κυρίω. Ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Γάλλοι επηρεάζονται τόσο άσχημα. Εμείς περνάμε λοιπόν τόσες πολλές περιφέρειες από νησί σε νησί περνάμε για να φτάσουμε στην υπηρετική Ευρώπη. Εμείς θα είμαστε οι πιο μειονεκτικοί και μην νομίζετε ότι εκλεγμένοι ω ως αιρετοί εκπρόσωποι δεν μπορείτε να καθυστερήσετε το πακέτο με κινητικότητα. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να καθυστερήσουν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αισθανόμαστε ότι μιλάτε από το βάθος της καρδιάς σας με πάθος. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα και να ανταποκριθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που γίνανε. Τις επόμενες εβδομάδες οι περισσότερες αποφάσεις θα περάσουν από το πολιτικό τμήμα στο πιο εμπορικό, αν θέλετε, τμήμα γιατί αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε συμβάσεις, εγκρίνονται συμβάσεις στο εμπορικό επίπεδο και θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν στο μέλλον και θα επηρεάσουν είτε το θέλουμε είτε όχι στο δεύτερο τμήμα, τρίμηνο με συγχωρείτε του 2019, τον τρόπο που θα διεξάγεται πλέον το εμπόριο. Και η δική μου ένωση και οι άλλες ενώσεις έρχονται σε επαφή μεταξύ τους για να δουν τελικά πώς θα δημορφωθούν οι τιμές μετά το Brexit. Αν οι πολιτικοί δεν μπορούν να μας δώσουν κάποιες αποφάσεις, τότε εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές μόνοι μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τελικά οι αποφάσεις θα ληφθούν στο εμπορικό το πλαίσιο, ακριβώ επειδή οι επιχειρήσει θα θέλουν να συνεχίσουν να μπορούν να λειτουργούν, θα θέλουν να μπορούν να εξυπηρετούν του πελάτε του και να διακινούν τα εμπορεύματά του. Επομένω, αυτά τα σχέδια έκτακτη ανάγκη, η προληπτική μα δράση, το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Τέιλορ. Σαφώς χρειαζόμαστε μια ασφάλεια, μια βεβαιότητα και μια προβλεψιμότητα. Αλλά ως επιχειρήσεις θα πρέπει να εργαστούμε με το χειρότερο δυνατό προβλεπόμενο σενάριο, το οποίο θα είναι το hard Brexit. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα αλλά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει να κάνουν και τις απαραίτητες επενδύσεις για να προσλάβουν προσωπικό που θα είναι σε θέση να διεξάγουν όλες τις νέες αυτές ε, διαδικασίες που θα πρέπει να επιβληθούν. Αυτό θα είναι πραγματική τραγωδία βέβαια να συμβεί. Θα είναι τεράστια απώλεια χρημάτων, αλλά θα είναι η πιο λογική επιχειρηματική απόφαση που μπορούμε να πάρουμε δεδομένων των κινδύνων και δεδομένων, δεδομένης αβεβαιότητας. Θα έλεγα λοιπόν προς τους ε, ευρωβουλευτές ότι ή δυνατόν θα πρέπει να περιμένουν να δούνε τι θα αποφασιστεί στις 14-15 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουμε να μπούμε μετά σε πιο σοβαρές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία που θα καλύψει όλα τα ζητήματα που δείξαμε σήμερα το πρωί. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να σωματωθούν όσον αφορά τα προσόντα, των οδηγών και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στην κυρία Φώστρα. εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Θεωρούμε πάντως ότι υπάρχει υφίσταται το ζήτημα αυτό της αναγνώρισης των προσόντων και νομίζω ότι μέσα σε όλες αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια εμπορική συμφωνία έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό το ζήτημα της αναγνώρισης των προσόντων και της αναγνώρισης της άδεια των οχημάτων καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος, είναι εντελώς άσκοπο να έχουμε μια εμπορική συμφωνία αν δεν υπάρχει, αν δεν εξακολουθήσει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και αμοιβαία αναγνώριση των αδειών των οχημάτων. Και προφανώς δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε αυτή τη στιγμή στη διαχείριση των συνόρων που είχαμε πριν από το 1992. Και ξέρετε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα επηρεαστούν από το Brexit, όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμεί έχουμε συντάξει το φυλάδιο αυτό το οποίο βλέπετε, όπου έχουμε 10 σημαντικά σημεία τα οποία πιστεύουμε θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να αποφύγουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και δεν αναφέρομαι σε κάτι νέο αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύονται ε, εμπορικές συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την απρόσκοπτη διέλευση των εμπορευμάτων όπως ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή και με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κέρν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να είμαι σύντομος στην παρέμβασή μου. Νομίζω ότι αυτά που ανέφεραν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές ε, με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό. Να αναφερθώ σε τρία σημεία όμως. Πρώτον, ένα ερώτημα που έθεσε ο κύριος Τέιλορ τι διακανονισμούς ε, χρειάζεστε σε τελωνιακό επίπεδο μετά το Brexit. Είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για τον κλάδο είναι όποτε λαμβάνει η χώρα η εκαθάριση, περνάει από το τελωνίο, τελωνίζεται, εν ένα φορτηγό, αυτό να γίνεται στο εσωτερικό της χώρας, όχι στα σύνορα διότι τα στοιχεία που μας έδωσε ο Τζέιμς προηγουμένως ε, σήμερα το πρωί ε, αν θέλουμε να έχουμε τέτοιους ε, ε τέτοιες διαδικασίες από ελληνική πλευράς ε, εάν γίνονται όλα αυτά στα σύνορα τότε οι ουρές θα είναι τεράστιες δεν θα μπορεί να ε, είναι η ροή, η ομαλή από την Ιρλανδία στο Μένο Βασίλειο. Και ένα θέμα τώρα που έδωσε ο κύριος Πίπερ για τα ψηφιακά σύνορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και αυτό εμείς το καλωσορίζουμε. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αξιολόγηση κινδύνου, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι σήμερα για να δούμε ε, πώς... Ε, ε, το φορτηγό και το εξοπλισμό του θα καθίσουν πιο ασφαλές ε, και βεβαίως ε, έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή και θα τη στηρίσουμε. Η τεχνολογία βεβαίως εξελίσσεται γρήγορα και αυτό αποτελεί πρόκληση για τον νομοθέτη διότι συχνά προχωράει πιο γρήγορα η τεχνολογία από την νομοθεσία και θα είναι μια πρόκληση για όλους να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, την κατάλληλη στιγμή ε, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο. Τώρα, εάν ε, υπάρχει αυτή η τεχνολογία, είναι διαθέσιμη στην αγορά, είναι προσβάσιμη στις τιμές, ε, προσιτές, εντάξει, αλλά δεν είναι μια απόφαση του κλάδου των οδικών μεταφορών να έχουμε αυτό ε, το, το, χωρισμό εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πότε σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Ήδη τώρα το Δεκέμβριο ε, θα πρέπει να είναι στο, στην πρώτη γραμμή της ατζένας των πραγματεύσεων το θέμα των δικών μεταφορών, διότι όπως είπε και ο Τζέιμς, ε, μπορεί να έχουμε πολλές συμφωνίες για διάφορα προϊόντα, για ε, διάφορους τομείς. Αν αυτά τα προϊόντα όμως δεν μπορέσουν να μεταφερθούν ε, έγκαιρα προς τους πελάτες, προς τους καταναλωτές, ε, τότε όλες αυτές οι συμφωνίες πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. Χάρτινη τίγρης. Ε, σας ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες ε, απαντήσεις. Τώρα παρακαλώ στις παρεμβάσεις των βουλευτών στις επόμενες ερωτήσεις, δηλαδή ένα λεπτό για ερωτήσεις για να προλάβουμε ε, να έχουμε και το δεύτερο πάνελ. Μετά θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαγκίνες, την πρώτη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, ευχαριστώ και για την ακρόαση. Ε, δεν ξέρω και τι να ρωτήσω. Είναι τόσες πολλές όταν ήρθα εδώ ήθελα απλώς να, να δείξω την υποστήριξή μου προς το έργο σας και προς τη συναδέλφο, στη συνάδελφο την Βερόνα Μέρφη. Ε, πολύ να θεωρήσατε την παρέμβασή σας, ε, την παρέμβασή της ως μια συναισθηματική παρέμβαση. Και βεβαίως είναι συναισθηματική διότι υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία στην Ιρλανδία για την πρόσβαση στην αγορά και δεν πρέπει να δώσουμε απάντηση σε αυτή την ανησυχία ως ότου δούμε πρόοδο στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Το ερώτημά μου λοιπόν ε, είναι άλλο. Για τις επιχειρήσεις πότε αυτή η αβεβαιότητα ε, είναι πλέον ε, αβάσταχτη και πρέπει να πάρθουν αποφάσεις δύσκολες. Ε, δεν είμαι βέβαιη ότι υπάρχει ένα plan B. Δεν ξέρουμε και ποιο είναι το σημείο αφετηρίας σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εταιρική σχέση. Θέλουν να ξέρουν πάντως οι συνάδελφοι που δεν προέρχονται από την Ιρλανδία ότι υπάρχει πραγματικά αυτή αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο κλίμα αβεβαιότητα. Είμαστε μια μικρή χώρα, χρειαζόμαστε πρόσβαση στις αγορές γρήγορα. Πρέπει το παρόν σύστημα να διαφυλαχθεί και να μην ε, αλλοιωθεί σημαντικά. Ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες. Συνεχίζουμε. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στα αγγλικά θα παρέμβω. Θα είμαι σύντομη είπε η Μαρέη ότι είστε μια μικρή χώρα και χρειάζεστε εμπόριο. Συμφωνώ απολύτως. Έχω συναντήσει εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών της Ιρλανδίας. Το ερώτημά μου είναι απλό. Πρώτα απ' όλα γνωρίζετε τι θα κοστίσει για σας το Brexit ε, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και δεύτερον, λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσει μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών της Ιρλανδίας ε, και των λοιπών Υπουργείων ε, των χωρών της Ένωσης. Δεν, πρέπει να τιμωρθείτε εσείς αν θέλει το Βασίλειο να φύγει. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Ε, ευχαριστώ η κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό που το πάνελ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό της μεταφοράς ε, αντίθετα με αυτά που λέει η κυρία Φώστερ εγώ δεν δέχομαι το γεγονός ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι όλα τα, όλες τις προδιαγραφές θα εφαρμοστούν διάφοροι συντηρητικοί ε, ε, πολιτικοί ε, υψηλόβαθμοι μας λένε το αντίθετο. Ο κύριος, ο κύριος Duncan Smith πρώην υπουργός εξωτερικών είπε ότι όταν ολοκληρωθεί το Brexit το 2019 πρέπει να προετοιμάσουμε μια αναθεώρηση ε, των ρυθμίσεων και πώς αυτέ αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών μας και τις επιχειρήσεις. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει νομικώς να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν θα ξέρω αν θα είναι μια βερσιόν της ελβετικής ε, συμφωνίας που θα λέει ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια και τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να συμπεριφυλαχθούν. Θα πρέπει να προτεραιότητα πάντως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μισελ Μπαρνιέ το είπε αυτό και ε, ε, θα ήθελα αυτό να γίνει σεβαστό. Μιλάμε για τις δεξιότητες, τις αδειοδότηση, τις ώρες εργασίας, ε, όχι με την έννοια τη επιβάρυνση. Θέλουμε να υπάρχουν ίσες συνθήκες. Λοιπόν, θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας από αυτού, διότι πρέπει απαραίτητο τα πράγματα να είναι σαφή, είτε σε μια συμπορική συμφωνία, είτε σε μια διμερή συμφωνία, είτε μια, ένας διακονισμός τύπου Νορβηγίας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άντερσον. Ο κύριος Βάνταλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ε, δυστυχώς, ε, λυπάμαι για το Brexit και κάπου ελπίζω ε, βαθιά μέσα μου να μην προχωρήσει. Αν προχωρήσει, ανέλπιστα, να μην είναι σκληρό Brexit, γιατί αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο με τις μεταφορές θα πληχθούν τόσο πολλοί τομείς και οι αεροπορικές μεταφορές, η αλληλεία και ούτω καθεξής όλοι. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω προς την ε, κυρία Μέρφη και στον κύριο Κέρνη. Καταρχάς, ε, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις ε, οι οποίες ενδεχομένως δεν ξέρω, υπάρχουν μηνύματα μήπως οι Ιρλανδικές επιχειρήσεις σκοπεύουν να μετακομίσουν στην υπηρετική Ευρώπη και κατά δεύτερον μιλάτε για την τέλεια θύελα που αναμένεται. Υπάρχει οποιοδήποτε θετικό σημείο όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Λούκα Σένσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε ότι το Brexit δεν συνεπάγεται μόνο κόστος για τις επιχειρήσεις μεταφορών, γιατί και το θέμα είναι και η πρόσβαση προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών ε, στις ε, ε, συναλλαγές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι οχταπλάσια σε σχέση με τον Καναδά. Μιλάμε για τεράστιο όγκο και αυτό θα προκαλέσει διοικητικά προβλήματα. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Τι κόστος θα προκύψει για τις επιχειρήσεις μεταφορών και για τους καταναλωτές λόγω των εξέλιξεων αυτών. Το δεύτερο θέμα. Στο Κοινοβούλιο κοιτάμε στην παρούσα φάση το πακέτο κινητικότητα και οι βουλευτέ ε, του ΕΒ Βασιλείου είναι πολύ δραστηροί. Πιστεύετε κυρίε και κύριοι ότι οι νέε αρχέ για καμποτάζ στι διεθνεί ε, μεταφορέ, για την ε, αναγνώριση των ικανοτήτων, για τα κοινωνικά ζητήματα, θα έπρεπε να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά τον Brexit και κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Επόμενος ομιλητής. Ε. Τρία σχόλια και μία παρατηρήσει σε ένα λεπτό το Brexit. Ξέρετε, δεν είναι φυσική καταστροφή, είναι μία απόρρια της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερη παρατηρήση. Οι συνέπειες είναι πολύ ασύμμετρε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό νομίζω ότι εξηγεί και την εφαρμογή ε, την διαφορετική εφαρμογή των ε, θεμάτων αυτών και τρίτον ότι η πολιτική εφαρμογή δεν έχει να κάνει με την γενικότερη πολιτική και θα έχουμε μεγάλε δυσκολίε Και μία ερώτηση λοιπόν έχω να σα κάνω γιατί έχω μόνο λεπτό στη διαθεσή μου. Οι τρεις παρεμβαίνοντες ε, πιστεύουν ότι υπάρχουν και πλέον εκτίματα σε ό,τι αφορά το Brexit. Ο den Kamp. Ε, έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Εγώ είμαι σε αυτή τη μικρή μειοψηφία που ακόμα δεν πιστεύω ότι θα γίνει καν το Brexit. Ε, για λύπηση βέβαια είμαι, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ίσως να υπάρχει ελπίδα. Η πιο σημαντική ερώτηση που έχω να απευθύνει προς τον κύριο Χουκάν είναι η εξή. Κάνατε καθόλου λόμπι ακόμα κατά του Brexit στην ε, Βρετανική κυβέρνηση και κατά δεύτερον, μήπως θα πρέπει να βρούμε τη λύση σε μια μακρά μεταβατική περίοδο, η οποία ενδεχομένως να μειώσει την πολιτική ζημιά, την οποία βλέπουμε εμείς ως Και μια ερώτηση, μια παρατηρήση μάλλον προς την κυρία Μέρφη. Ε, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μακίνης ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε την Ιρλανδία. Αλλά το να αναβάλουμε το πακέτο κινητικότητα λόγω του Brexit θεωρώ ότι θα αποτελούσε διπλή ζημιά για μας και το βρίσκω απαράδεκτο ως λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φαντακάμπλε, η πρόεδρος, ο κύριος Κράμερ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Υπάρχουν σχέσεις ε, με την Νορβηγία, με την Ελβετία, με τρίτες ε, χώρες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το υποστηρίζεται αυτό ως προσέγγιση, γιατί αυτό δεν θα προκύψει επειδή θέλει να εξοικονομήσει χρήματα το Ηνωμένο Βασίλειο. Α, έχει και πλανεκτήματα η λύση αυτή. Θέλετε λοιπόν από πλευρά της χώρας σας να περάσει κάτι τέτοιο. Να τύχει δηλαδή ίδια αντιμετώπιση και το Ηνωμένο Βασίλειο των εξάρτητων τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η Ελβετία και στην Αρβηγία. Και τέλο, τι γίνεται με τη μάχη, με το τούνελ τη μάχη. Έχετε κάποια ιδέα και τι θα υποστηρίζετε ω λύση. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Είδατε πόσε είναι οι ερωτήσει. Και μάλιστα ερωτήσεις ε, όπως για παράδειγμα αυτή της κυρίας Μαγκίνες, που ακριβώς βασίζεται σε αυτές τις ε, ανησυχίες. Ε, αυτό που ρωτάει είναι... για να υπάρχει ένας, ε, ένα σχέδιο, αν θέλετε, από πλευρά του κλάδου, του οικονομικού. Και επίσης, πολλές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το κόστος. Πώς θα μας κοστίσει πια αυτό το Brexit. και για τους μεταφορείς. Και να αναφέρω και την ερώτηση του κυρίου Ρίκε. Έχει και κανένα πλεονέκτημα τελικά αυτό το Brexit. Και όπως είπε και ο κύριος Φόντεν Κάμπε, που δεν το πιστεύει ότι θα γίνει. Υπάρχει καθόλου και αυτή η αίσθηση στον δικό σας τον κλάδο. Ότι δεν θα γίνει δηλαδή. Είναι σημαντικές προφανώς οι ερωτήσεις. Και δίνω το λόγο στην κυρία Μέρφυ για δύο λεπτά. Thank you. thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάλι όλους όσοι πήραν το λόγο. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Μαρέ Μαγκίνες, η οποία πραγματικά είναι πολύ καλή φίλη των, της Ένωσής μας και των Ιρλανδών οδηγών εμπορικών μεταφορών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Μαγκίνες και τους υπόλοιπους που πήραν το λόγο. Να απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση της Μαρέιντ. Το Brexit για τους Ιρλανδούς οδηγούς, τους Ιρλανδούς επιχειρηματίες, ουσιαστικά προφανώς θα είναι αρνητικό. Ξέρετε ότι οι έξι κομιτείες της Βόρειας Ιρλανδίας μπορούν να εργάζονται, μάλλον θα έχουν ένα έλλειμμα της τάξης του 20%. Τα προβλήματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ήδη το έλλειμμα αυτό έχει προκύψει. Το 20% του κλάδου αυτού οδικών εμπορευματικών μεταφορών έχει ήδη επηρεαστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, που μας δανείζουν δηλαδή, που ανησυχούν για την εξέλιξη των πραγμάτων. Εμείς ε, προφανώς προχωρούμε σε διαβούλευση, είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία και τα Υπουργεία μας είναι σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία του Ηνωμένου Βασιλείου και εξετάζουμε όλες τις συναλλακτικές ήδη από το 2017 είχαμε εκτιμήσει σε 200 εκατομμύρια το κόστος από το Brexit, μόνο και μόνο από τις καθυστερήσεις. Εγώ πραγματικά, αν πρέπει να επομιστώ το κόστος αυτό, θα βρεθώ εκτός εργασίας πραγματικά. Τέσσερα φορτηγά έχω, μια μικρομεσαία επιχείρηση μου σαστικά με τα τέσσερα αυτά φορτηγά τα οποία δεν μπορώ να καλύψω πλήρως συνεχώς με οδηγούς θα χάσω πάρα πάρα πολλά χρήματα και ήδη πληρώνω περί τα πάνω από χίλια ευρώ σε φόρους. Και βέβαια δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση να μετακινήσω την επιχείρησή μου σε ένα άλλο κράτο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την πίεση αυτή θα αρχίσουν να έχουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω επιπλέον επιζήμιο παράγοντα έχουμε και την αρνητική πλέον συναλλαγματική ισοτιμία. Καταλαβαίνετε ότι διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρώ ότι οι πρακτικές που υφίστανται αυτή τη στιγμή, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές δεν θα γίνουν αναγκαστικά πιο αυστηρά. Θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά το Brexit. Πάλι απαντώ σε μια ερώτηση του κυρίου Βαντάλεν. Εγώ έχοντας μια μικρή τελικά επιχείρηση δεν θα καταφέρω τελικά να πάω σε μια άλλη χώρα. Πώς θα καταφέρω τελικά να μεταφράσω μόνο και μόνο σε πέντε διαφορετικέ γλώσσε τη σύμβαση την οποία συνάπτω με τους οδηγούς μου καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ως υποχρέωση αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να προχωρώ ουσιαστικά στις μεταφράσεις αυτές μετά το Brexit. Πού θα βρω τους μεταφράστες, πώς θα καταφέρω τελικά να πληρώσω τις μεταφράσεις αυτές, ακόμα και αν πάω στις πρεσβείες μας, νομίζω ότι θα πρέπει να πληρώνω 200 ευρώ τη μετάφραση. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι δαπάνες και όλες αυτές οι νέες διοικητικές ρυθμίσεις αρχίζουν και επιβαρύνουν πάρα πολύ την εργασία μας και πολύ φοβάμαι ότι η γραφειοκρατία θα αυξηθεί. Και το ερώτημα το οποίο θέτουμε μετά το δημοψήφισμα για το Brexit είναι πραγματικά για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση και πραγματικά θα απομακρυνθούμε εμεί ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε φορά που μακρινόμαστε, ζημιωνόμαστε και χρηματικά. Αυτή είναι η προοπτική, αν θέλετε, της Ιρλανδίας. Σα ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Χούκαμ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Μέρφη. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε τελικά τι γίνεται με το ζήτημα της νομοθεσίας. Έχουμε έρθει σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία και προσπαθούμε να καλύψουμε όλο τον κλάδο και των εμπορευματικών μεταφορών και των υπόλοιπων οδικών μεταφορών, προκειμένου να έχουμε και στο μέλλον ένα βιώσιμο και ασφαλές σύστημα μεταφορών. Και μολονότι είχαμε ασχοληθεί με τους κανονισμούς και τις οδηγίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εγκρίθηκαν και για τη δική μου τη χώρα, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάποιοι από τους κανονισμούς αυτούς θα υφίστανται και στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι ε, μετά το Brexit ε, θα πρέπει να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Τώρα το κόστος εξαρτάται από το πόσο σκληρό θα είναι το Brexit. Ποια θα είναι οι νέοι διακανονισμοί όσον αφορά τα νέα σύνορα. Ξέρετε ότι ένα φορτηγό το οποίο κάθεται ένα λεπτό σε μια ουρά του στοιχίζει περίπου μία λίρα. Μία λίρα το λεπτό είναι ο κόστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν πάρουμε όλε τι καθυστερήσει που θα προκύψουν και όλα τα φορτηγά που θα περιμένουν σε ουρέ, τα ποσά θα είναι τεράστια. Επιθυμούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία του Brexit. Ξέρετε ότι η επιχειρηματική κοινότητα και ιδίω ο δικό μα ο κλάδο αναγνωρίζει αυτό το υπόθηκε πριν από λίγο απεφάνθη ο Βρετανικός λαός, δεν είναι κάτι το οποίο ζήτησε αναγκαστικά ο δικός μας ο κλάδος, πάντως δεν εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες και λέμε με κάθε δυνατή ευκαιρία ποιες θα είναι οι δεινές επιπτώσεις, ιδίως ενός σκληρού Brexit όσον αφορά τις ε, οδικές εμπορευματικές μεταφορές και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα γενικότερα του τομέα μεταφορών και στον Ηνωμένο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, Υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα από τον Brexit. Υπάρχουν. Γιατί δεν νομίζω ότι η δική μου η Ένωση Οδικών Μεταφορών θα είχε ποτέ τη δυνατότητα να έρθει και να μιλήσει εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας τι καταπληκτική εργασία κάνουμε προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη ροή μεταφορών και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευκαιρία αυτή δεν θα μας είχε δοθεί αν δεν είχε προκύψει το Brexit. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μια θετική εντό αγωγικών επίπτωση είναι ότι στη συζήτηση αυτή που γίνεται για το Brexit, αν μη τι άλλο, προβάλλεται λίγο περισσότερο και ο δικό μα ο ρόλο σε εσά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο ομιλητή ο κύριο Ντάνιελ Κέρν. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Ρικέ, αν υπάρχουν πλεονεκτήματα τα οποία να απορρέουν από το Brexit. Κοιτάξτε, τα μέλη της IRU τη Διεθνού Ένωση Οδικών Μεταφορών πρέπει να σας πω ότι ανησυχούν. Υπάρχει πολύ μεγάλη βεβαιότητα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ιδίω εξαιτία του πολύ αργού ρυθμού με τον οποίο κινούνται οι διαπραγματεύσει μέχρι στιγμή. Αυτό μα προκαλεί πολλέ ανησυχίε. Μέχρι στιγμή δεν μπορούμε να δούμε πλέον εκτίματα από τον Brexit όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μα τον επαγγελματικό κλάδο. Πρώτον αυτό. Τώρα, κύριε Λουκασένσκα, έθεσε ένα ερώτημα για το καμποτάζ. Αν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά το Brexit, κοιτάξτε, οι κανόνες περί καμποτάζ, όπως τους ξέρουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύουν για τρίτες χώρες. Οτιδήποτε λοιπόν ε, αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας με τους Βρετανούς θα είναι αντικείμενο μιας ε, ξεχωριστής συμφωνίας στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει να υπάρχουν επίσης δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τις άδειε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μορφή θα πάρει αυτή η μελλοντική συμφωνία τώρα όσον αφορά τις επιχειρήσεις θα μετεκατασταθούν οι επιχειρήσεις μας. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις εμπορικών οδικών μεταφορών διαφέρουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αν κάποιος είναι, αν θέλετε, βαθιά ριζωμένο στα πλαίσια μιας κοινότητας, στα πλαίσια μιας χώρας ή περιοχής, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά μία νυχτή να μετακατασταθεί σε μία άλλη εταιρεία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ακριβώς τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μία άλλη οποιαδήποτε παραγωγική επιχείρηση που κατασκευάζει προϊόντα η οποία πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα. Δεν ζητάμε δεύτερο δημοψήφισμα, δεχόμαστε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα του πρώτου δημοψηφίσματος, αλλά μη τι άλλο θα θέλαμε να έχουμε διευκόλυνση του εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και μετά το Brexit, προσπαθώντας να μετριάσουμε στο βαθμό του δυνατού τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Πρόεδρος, κυρία Μάρφη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα απλώ να πω ότι το μόνο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε εκ νέου duty free. Αυτό είναι το μόνο πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να προκύψει από το Brexit. Πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίε του πρώτου πάνελ. Α χειροκροτήσουμε του παρεμβαίνοντε, του καλεσμένου μα. Σα ευχαριστώ πραγματικά ειλικρινά για την ποιότητα των παρεμβάσεών σα, για την εμπειρογνωμοσύνη σα αυτή γιατί ότι μας είπατε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένα πλεονέκτημα στο Brexit, ήσασταν απόλυτα σαφείς διαγράψατε ένα μελλοντικό σενάριο το οποίο διέπεται από αβεβαιότητα και πάρα πολλές ανησυχίες. Κάντε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Μας είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές αυξήσεις, τελειωνιακές και άλλες, διοικητικής φύσης, ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι διοικητικοί έλεγχοι, κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα προκύψει από τα πάρα πολλά φορτηγά που θα περιμένουν στα σύνορα και το καθεξής. Μην ανησυχείτε και εμείς εκ του σύνεγγης παρακολουθούμε την πορεία διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν πρέπει να κάνουμε όμως τίποτα διότι θεωρούμε και εμείς ότι καθυστερούν πάρα πολλοί διαπραγματεύσεις. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση διαπραγματεύσεων, προσπαθούμε να το προετοιμάσουμε τη δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ στην Επιτροπή μας να έρχεστε να μας βλέπετε και να μας ενημερώνετε για τα του κλάδου σας. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους καλεσμένους μας στο δεύτερο πάνελ να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Προχωράμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Πάντα όσον αφορά τις μεταφορές, αλλά αυτή τη φορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, με τους θηροδρόμους. Και είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκονται εδώ κοντά μου άνθρωποι που γνωρίζουμε αρκετά καλά. Πρώτα ο Ζακ Γκουνό, ο διευθυντής, κλασικός διευθυντής του, Euro, του ε, σας ευχαριστούμε. Ο Λίμπορ Λόχμαν, εκκλησικός διευθυντής του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιδροδρόμων. Ε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Και βεβαίως η Λόρα Ράιτ, η εκπρόσωπος του Rail Delivery Group, το θέμα των ε, ε, εμπορευμάτων που είναι σημαντικό ζήτημα. Όπως και με το πρώτο πάνελ θα έχετε 7 λεπτά για να μας πείτε πώς εσείς βλέπετε τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Μένου Βασιλείου στον κλάδο σας και πώς θα θέλατε η Επιτροπή Μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, ε, να κινηθεί έτσι ώστε να μην είναι μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Είδαμε πάντως στις οδικές μεταφορές τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια πανευθερής κατάσταση και στις, στις, ε, ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Ράιτ, 7 λεπτά. Um, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι η Λόρα Ράιτ, είμαι επικεφαλής της διεθνούς πολιτικής του Rail Delivery Group. Ο στόχος μας είναι οι βρετανικές υποδομές ε, και οι εταιρείε μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών να συντονίζονται για να βελτιώσουν τι υπηρεσίε του. Είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα. 240.000 άνθρωποι εργάζονται στι ε, ε, συνδρομικέ μεταφορέ. Ε, εκατομμύρια άνθρωποι μεταφέρονται. 65 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο σε εμπορεύματα και αυτά τα στοιχεία βεβαίως είναι γνωστά στα, στα κράτη-μέλη της Ένωσης εισαγωγές, εξαγωγές αγαθών, υπηρεσιών, ε, μεταφέρονται άνθρωποι, είναι και η μόνη σύνδεση ε, με, το, με την υπηρετική Ευρώπη, η, η χερσαία μεταφορά, ε, ως χερσαία μεταφορά δηλαδή, ε, και έχουμε τρεις προτεραιότητες ό,τι αφορά τις για το Brexit. Πρώτα, αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά, ε, ομαλή διασυνοριακή διέλευση και ε, οι θέσει απασχόληση του τομέα. Πρώτα, πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, εμεί θεωρούμε ότι εδώ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στην, στην Επιτροπή Μεταφορών με το πακέτο για την κινητικότητα, ανοίγουν οι αγορές, ε, καινοτομία, περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αργές καταναλωτές, ε, όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, ε, ε, επενδύσεις, απασχόληση προς την Αμένο Βασίλειο από τις εταιρείε αεροδρόμων. Πρέπει να μάθουμε από την επιτυχία μας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως αυξάνουν την παρουσία τους στην υπηρετική Ευρώπη και πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές για να μπορούμε να εξάγουμε και την πραγματομοσύνη μας. Χρειάζεται αμοιβαία λοιπόν ε, απρόβαση στην αγορά. Αυτό συζητείται σε πολύ ψηλό πολιτικό επίπεδο. Εμεί είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού ό,τι αφορά τι υπηρεσίε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, αλλά και ε, πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για την ομαλή διέλευση των συνόρων. το συζητήσαμε και το πρωί σήμερα για τι χερσαίε μεταφορέ. Όμω για μα το, το τον κάτω από τη μάχη είναι ένα πολύ, βασ, μια πολύ, ένα πολύ βασικό σημείο διέλευση μεταξύ του Βασιλείου και Περιοχή Ευρώπη. Είναι ένα κρίσιμο σύνδεσμο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου, ακόμα και όταν το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί είναι τρίτη χώρα. Το να μπορεί να ταξιδέψει κάποιο από το τούνελ αυτό ε, θα πρέπει να. Ε, ε, τα τεχνικέ προδιαγραφέ να είναι εγκεκριμένε και από την Βασιλεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία τα, οι προδιαγραφές αυτές και να μπορούμε να δράσουμε ε, και να εμπορευτούμε υπηρετικά στο Βέλγιο, στη Γαλλία και αλλού. Ε, οι διαχειριστές υποδομών στις διασυνοριακές ε, οδούς, εφόσον αλλάξουν ε, τα στοιχεία συμβατότητας, θα πρέπει... Ναι, μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο αργά. Ναι, συγγνώμη, δεν περνάνε πολύ καλά μεταφραστέ. φαντάζομαι, λέει ο Μιλήτρια. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόθεση από τις επιχειρήσεις ή από του διαχειριστές υποδομών σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή διέλευση να αλλάξουν οι κανόνες συμβατότητα. Ε, πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των αδειών για του μηχανοδηγού. Δεν ξέρουμε βεβαίω ε, τι ακριβώ θα γίνει με τον Brexit. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε ένα σενάριο όπου δεν θα υπάρχει αμοιβή αναγνώριση των αδειών ε, εκμετάλλευσης, ε, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολε δύσκολες οι επιχειρήσεις μας. Χωρίς αμοιβή αναγνώριση, παραδείγματος χάρη των, ε, διπλωμάτων οδήγηση, θα πρέπει κάποιος να έχει δύο διπλώματα ή να αλλάζουμε οδηγό στα σύνορα. Ε, Όμω με συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και κυβερνήσεων θα μπορούσαμε, να βρούμε μια λύση. Η συμμετοχή στην Τελωνιακή Ένωση της, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να, μας επιτρέπει να εισάγουμε και να εξάγουμε χωρί να υπάρχει δήλωση για, για τους ε, κανόνες προέλευσης, ε, ε δεν χρειάζονται περισσότερη έλεγχη για την ασφάλεια και αυτό έχει λιγότερε καθυστερήσει. Αυτό θα έχει λοιπόν επιπτώσει. Ε, ε, υπάρχει μια απλουστευμένη διαδικασία για τα αγαθά και όλα τα αγαθά που περνούν από το τούνελ εκπροσωπούν το 1 τέταρτο του εμπορίου μεταξύ της Ευρώπης 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, χωρίς ε, σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και στους τελωνιακούς υπαλλήλου και την τεχνολογία όπως τα σκάνερ ε, θα είναι πραγματικά δύσκολο να υπάρξουν επιπτώσεις στα γαλλικά αλλά και στα βρετανικά σεοδρομικά δίκτυα. Αυτό θα έχει βεβαίως επιπτώσεις και σε άλλα σεοδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη. Για τους ανθρώπους τώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι ταλαντούχοι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη. Ε, είναι χιλιάδες, ε, περίπου χίλιοι άνθρωποι που εργάζονται στο σιδηρόδρομο από την Ευρώπη. Πολλοί, ε, πολλές ε, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στον τομέα της προσφοράς παροχής υπηρεσιών, ε, εργάζονται για τρει μήνες αλλά και για πολλά χρόνια ορισμένε φορέ. Πρέπει να παραμείνει αυτή η δυνατότητα ε, αποσπασμένων εργαζόμενων, ε, ε, πολλοί εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν το τούνελ κάτω από τη μάχη προέρχονται από πολλές εθνικότητες, έχουν τις δεξιότητές τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια λύση με μια σωστή σχέση κόστους ωφέλους η Ευρώπη των 27 βασίζεται και στην ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ υπηκών Ευρωπαίων και Βρετανών και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια κοινών project. Παραδείγματο χάρη το Crossrail που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών. Εκεί δουλεύουν πάνω από 50.000 εργαζόμενοι, οπότε υπάρχει, να υπάρχει το 2009, εκτιμά, περίπου 5% των συνεργειακών αποσχολούμενων είναι Ευρωπαίοι ε, υπηκόοι όλοι αυτοί έχουν γνώσει, έχουν δεξιότητε από αυτό το project και μπορούν να τα μεταφέρουν σε άλλε σημαντικέ ε, project υποδομών στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ε, το, την, ε, το εργατικό δυναμικό το οποίο είναι καταρτισμένο για να μαθαίνουμε. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό για τις σιρόδρομο, όχι μόνο για να έχουμε ανταγωνιστική αγορά, αλλά και να μπορούμε να μοιραστούμε τη, τη, μοναδική αυτή εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Συμπερασματικά λοιπόν, οι σειρόδρομοι του Μένου Βασιλείου δεσμεύονται να συνεργαστούν με τι με τις Βρυξέλλε, με την Βρετανική κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την διαδικασία αποχώρηση του Μένου Βασιλείου. Πρέπει αυτά τα σχέδια να υποστηρίξουν τον ευρωπαϊκό Σειροδρομικό χώρο ε, και ε, να υπάρξουν ωφέλη για του επιβάτε αλλά και για τι μεταφορέ. Δεν ξέρω αν ήμουν πολύ γρήγορη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε. Με τον Λόχμαν. Για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ ο ρόλος μου να μιλήσω μετά την συνάδελφο ή μετά τις ανησυχίες που ξέρουμε ότι υπάρχουν στον τομέα των δρόμων και τα θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα μας πραγματικά. Σε πρώτη φάση, το CR, όπως θα ξέρετε, εκπροσωπεί την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που κινούνται σε ευρωπαϊκές τροχές και στην Υπηρετική Ευρώπη αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία και εκπροσωπούμε, αντιπροσωπεύουμε τα συμφέροντά του ε, στι Βρυξέλλε. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία ανησυχία μα, Καταρχά, χάρη σε εσά και στι προσπάθειέ σα στο παρελθόν, καταφέραμε πρόσφατα να ιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Περιοχή, τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Τομέα και Χώρο. Θέλουμε προφανώς, να επεκταθούμε και προς την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, αυτά που έχουμε πετύχει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό για μας... Ε, είναι ο στόχος μας σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Η νομική βεβαιότητα λοιπόν για τις επιχειρήσεις η οποία θα είναι δυνατή και θα πρέπει να, εγγυηθούμε και για μετά το Brexit. Πρόσβαση στην αγορά δεν πρόκειται να ε, επαναλάβω αυτά που είπε η συνάδελφο. Ω τμήμα τη νομοθεσία προβλέπεται αμοιβαία πρόσβαση στι αγορέ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Υπηρετική Ευρώπη. Θέλουμε αυτό να συνεχιστεί προφανώ. Αυτό θα ήταν αποφελές και για τους πελάτες και για τους επιβάτες και αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δευτερευρωθεί. Μιας και μιλάμε και για επιβάτες σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμβάσεις, σε ό,τι αφορά όλες τις συμβάσεις. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πρόσβαση προκειμένου να υπάρχει και καλή συνεργασία μεταξύ των ομοφοδικών αρχών και από τις δύο πλευρές της μάχης. Η κινητικότητα του προσωπικού. Τι να προσθέσω πέρα από αυτά που είπαν συνάδελφοι για τις οδικέ μεταφορές. Ε, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει κινητικότητα των ατόμων για να υπάρξει όφελος ε, από το ταλέντο, από την γνώση, από την προγνωμοσύνη όλων. Ιδάλλως θα πληχθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο απλά επαναλαμβάνει τα όσα έχουμε ήδη ακούσει. Τεχνικοί κανόνες τώρα, για να τους κοιτάξουμε πιο εντελεχώς. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή του ε, Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου για την υλοποίηση και τη μεταφορά των οδηγιών για την λειτουργικότητα και την ασφάλεια για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνδροδρόμων. Και από την άλλη υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο θα ορθωθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο θα παρεμποδίσει την λειτουργία μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν από τεχνική άποψη ε, τι θα γίνει. Ό,τι γίνει από τεχνική άποψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνει, να βρει αντίκρισμα και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό θα έχει να κάνει και με την αναγνώριση των σχετικών ε, εγκρίσεων και αδειών και θα πρέπει επίση αυτό να εξασφαλίσει καλή συνεργασία στο μέλλον μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλεία σε ό,τι αφορά α, και την επικοινωνία μέσω τη Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία για του δρόμου και σε ό,τι αφορά και του ε, ε, εμπειρογνώμονε που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις τον τεχνικό κανονισμό και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι απόφευκτο. Ιδάλλως, ό,τι έχουμε κάνει τις τελευταίες δύο δεκαετίες θα τα ξεκινήσουμε αυτό ξανά από την αρχή. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο είναι και στη δική σας ατζέντα από ό,τι μας παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, και το κινητικότητα σε ό,τι αφορά και την οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες θα είναι οι μελλοντικέ εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον διαλειτουργικό ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν οι σιδηροδρομοί να μείνουν σε εξίσου σημαντική θέση. Μη σα πω να ενισχυθεί και η σημασία του στο μέλλον, προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τελωνία και τα σύνορα, τι να προσθέσουμε από αυτά που μα είπαν και οι συνάδελφοι από τι οδικέ μεταφορέ μετά από όσα έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια για τα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας, ε, Βρεσιλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου και φυσικά και για το, τη σειρά της μάχης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις μας και να λειτουργούμε τις επιχειρήσεις μας χωρίς μεγάλες ε, εμπόδια και στρεβλώσεις. Αυτό θα ήταν καταστροφή έρευνα και ανάπτυξη. Και καινοτομία, συγγνώμη. Χρόνια πάλι μας πήρε να προσεγγίσουμε τα προγράμματά μας να γίνει αυτή η μετάβαση. Και πραγματικά βάζουμε πάρα πολλούς πόρους και προσπαθία και χρήματα στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τις αμοιβέ εισφορές προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει φυσικά να επιτρέψουμε στους εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν να συμμετέχουν όχι μόνο στην ψηφιοποίηση, αλλά και γενικότερα στον πιο ανταγωνιστικό ανταγωνιστική διαμορφωσή των, του κλάδου. Τέλος, βατικές ρυθμίσεις. Αν όλα αυτά που σας είπα καταφέρουμε να ισχύσουν για να μην διακοπεί η παροχή των υπηρεσιών και να υπάρχει πραγματικά ένας πραγματικά ευρωπαϊκός, ε, ευρωπαϊκός χώρος, θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση μέχρι ότου να δημιουργηθεί μια δημιουργή συμφωνία, να μην υπάρξει χάσμα, κενό νόμο μεταξύ αυτών που ισχύουν σήμερα και μεταξύ των μελλοντικών ε, διατάξεων που κανείς δεν τις γνωρίζει σίγουρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Κουνού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείστε με την σύραγγα της μάχης. Πρόκειται για ένα μοναδικό project. Δημιουργήθηκε από μια διεθνή συνθήκη πριν από 30 περίπου χρόνια. Πρόκειται για μια τεράστια καινοτομία προκειμένου το τούνελ κάνω από τη μάχη να έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το Brexit δεν μπορεί και δεν πρέπει να διακόψει την εύρυθμη αυτή λειτουργία του νομικού αυτού πλησίου. Καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ιδίως όταν βρισκόμαστε και τόσα μέτρα κάτω από τη μάχη. Πρόκειται για μια σιδεροδρομική και οδική διασύνδεση πάρα πολλών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά οχήματα και φορτηγά τα οποία επιβαίνουν σε αμαξοστοιχίες προκειμένου να περάσουν από τη μία πλευρά της, μάχη μάχης στην άλλη. Άρχισε να λειτουργεί το 1994 το Eurotunnel είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται, διαχειριζόταν μάλλον μέχρι το 1986 την διασύνδεση αυτή και έχουμε πάρα πολλούς που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς το Brexit θα επηρεάσει το Eurotunnel και γενικά τα κυκλοφορία στη σύραγγα της Μάνχης και θεωρώ ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την μεταφορική αυτή διασύνδεση με τη σύραγγα της Μάνχης και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα χερσαίο σύνορο. Μπορούμε να περάσουμε μέσω τη διασύνδεση αυτή τη χερσαίας από την υπηρετική Ευρώπη προς το Μένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρχουν χερσαία σύνορα δηλαδή μόνο μεταξύ τη Ιρλανδία και της Βορείου Ιρλανδία. Και κάτι πολύ σημαντικό που το βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, από τότε που άρχισε να λειτουργεί το τούνελ, έχουμε εκατοντάδε εκατομμύρια επιβατών, οχημάτων, εμπορευμάτων που διέσχισαν τη σύραγγα της μάχης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ζωτική σημασία το τούνελ αυτό. Όσον αφορά το 2016, όσον αφορά τα εμπορεύματα και την αξία των εμπορευμάτων 116 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν ουσιαστικά από τη σύραγγα της μάχης. Αυτό αντιστοιχεί περίπου 25% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Υπηρετικής Ευρώπης και έχει να κάνει με όλες τις χώρες της πυρωτικής Ευρώπης, γιατί ένα 62% των εξαγωγών της υπηρετικής Ευρώπης πηγαίνουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για τον Brexit, ένα δεύτερο μήνυμα. Αν τεθεί εν κινδύνο η σημαντική αυτή εμπορική ροή εμπορευμάτων μεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με πάρα πολλούς εμπόρους και πάρα πολλού επιβάτες, καθότι ένα 62% όπως είπαμε των εξαγωγών πηγαίνει προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνετε και θα ήθελα να πιστήσω σε αυτό την προσοχή των ευρωβουλευτών ότι θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες επιζήμιες επιπτώσεις από το Brexit όσον αφορά την εμπορική αυτή ροή, όσον αφορά την απασχόληση επίση. Καταλαβαίνω ότι οι επιπτώσει αυτέ ήταν σημαντικότατε όχι μόνο για το Βασίλειο αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε και δεν το λέμε αρκετά συχνά. Το Brexit και ουσιαστικά η λειτουργία τη έργα τη μάχη αφορούν πολύ περισσότερο, θα πρέπει να ανησυχούν πολύ περισσότερο την πυροτική Ευρώπη από ότι το Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να ασχοληθούμε και με το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον που χρησιμοποιούν από εμπορική και επιβατική πλευρά τη σύραγγα τη μάχη, καθότι οι ενέργειε μεταφορέ κοστίζουν πολύ πιο ακριβά. 100.000 φορτηγά, βαρέα φορτηγά σε καθημερινή βάση περνάνε από τη σύραγγα τη μάχη. Μέσα σε μία μέρα λοιπόν, κατά μέσο όρο, 100.000, 100 χιλιόμετρα μάλλον φορτηγών περνάνε από το σύρεκα της μάχης και φτάνουμε πολλές φορές στα 10.000 χιλιόμετρα, 200 λοιπόν χιλιόμετρα φορτηγών σε κατάσταση συνεχούς ροής περνάνε από τη σύρεκα της μάχης. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα εφόσον σας φαίνονται όντως εντυπωσιακά, θα πρέπει να έρθετε πραγματικά να δείτε πώς έχει γίνει η σύραγγα της μάχης. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Η παραμικρή αναστάτωση, η παραμικρή διακοπή της εύρυθμης αυτής ροής μεταφοράς δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα παραλύσει όχι μόνο τη Γερμανία αλλά και τις χώρες Μπενελούξ αλλά ακόμα και τη Γερμανία και γενικά όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που διοχετεύουν προϊόντα προς το Νομένο Βασίλειο. Παναλαμβάνω μεγαλύτερο το πρόβλημα για την πυρωτική Ευρώπη από ό,τι για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να απορροφήσουμε λοιπόν όλη αυτή την καθημερινή κυκλοφορία θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή εύρυθμη ροή της κυκλοφορίας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε σήμερα τα Γάλλο-Βρετανικά σύνορα, τα οποία έχουν μετακινηθεί ουσιαστικά στην γαλλική επικράτεια και πέρα γίνονται όλοι οι έλεγχοι, καταλαβαίνετε ότι μετά το Brexit θα επέλθουν αλλαγέ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμω να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα συστήματα πληροφορική που ισχύουν αυτή τη στιγμή στη γαλλική πλευρά, προκειμένου η ροή αυτή των επιβατών και των εμπορευμάτων να γίνεται απρόσκοπτα γιατί όπως σας είπα στην αντίθετη περίπτωση θα ζημιωθεί πάρα πολύ και η εμπορική ροή και τα οικονομικά λοιπόν αποτελέσματα, αλλά και ο τομέας απασχόλησης, αλλά και ο περιβαλλοντικός τομέας. Καταλαβαίνετε ότι η πτυχή αυτή περιβαλλοντική, καθώς επίσης και η πτυχή των διασυνδεδεμένων μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντική. Η μόνιμη αυτή ε, διασύνδεση μέσω της μάχης έχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, αντιστοιχεί ουσιαστικά στην αρχαισαίο σύνορο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν τον κανονισμό όπως ισχύει αυτή τη στιγμή ή το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως έχει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι θα μπορούσαμε να διηγηθούμε ακόμα και σε ατυχήματα, ακόμα και σε απώλεια ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το έχουμε κατά νου. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλους τους απαραίτητους πόρους της πληροφορικής που διαθέτουμε προκειμένου να μπορούμε να έχουμε γρήγορους τελωνιακούς ελέγχους. Θα πρέπει ακόμα και αν έχουμε τελικά τελωνιακούς ελέγχους να μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα συστήματα εκτελονισμού. Νομίζω ότι ε, αυτή την ευθύνη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού και θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβουν στα πλαίσια διαπραγματεύσεων και να πούνε στους διαπραγματευτές ότι ε, έχετε ένα 70% των εμπορικών ροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πηγαίνουν τελικά προς το Μένο Βασίλειο. Δεν μπορείτε λοιπόν σε καμία περίπτωση να στραφείτε κατά της καταπληκτικής αυτής επιτυχίας των τελευταίων 30 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι σαφές αυτό που μας είπατε να μην καταστρέψουμε αυτά που οικοδομήθηκαν με κοινή βούληση στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αυτό είναι το σαφές μήνυμα που μας στέλνετε. Είναι σαφής και η ανησυχία στα λόγια σας. Ευχαριστώ και από τις τρεις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στις επιπτώσεις ε, για το θέμα ε, της ε, ε, της απασχόλησης, για το θέμα των μεικτών μεταφορών, πώς θα αλλάξει η νομοθεσία. Ε, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε δύο τις νομοθεσίες, δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εάν ξεκινήσουμε από την αρχή. Επίσης δώσατε και κάποια στοιχεία αριθμητικά, εξαιρετικά, ε, εμπεριπωσιακά, 240.000 άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα αυτό, τι θα γίνει με αυτούς. 41.000 Ευρωπαίοι εργαζόμενοι ε, τι θα γίνεται, ξαναδούμε την νομοθεσία ε, και επίσης ε, είπατε ότι είναι κάτι που λειτουργεί καλά τώρα ε, ο σύνδεση με τον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί να καταστρέψουμε κάτι έτσι βία, κάτι που λειτουργεί τόσο καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση ο κύριος Πίπερ και πάλι έχει το λόγο παρακαλώ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Δεν θα χρειαστώ καν τα δύο λεπτά. Γιατί τα στοιχεία αυτά ήταν τόσο ξεκαθαρά. Και δεν πιστεύω ότι οι άδειε για τους ε, οδηγούς σιδηροδρόμων και ούτω καθεξής ε, στο πακετό συνδρομικών μεταφορών. Όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία θα πρέπει να τα θίξουμε γιατί μπορεί κάτι να βγει από το πακέτο. Η πολιτική μου εμπειρία μου λέει ότι καλό θα ήταν να τα κοιτάξουμε όλα αυτά από κοινού. Κάπως όμως ε, υπερβάλλουμε το να λέμε δηλαδή ότι στο, στη Σιράγκα ενδεχομένω να υπάρχει άλλη νομοθεσία και αυτό να οδηγήσει σε καταστροφή. Σας παρακαλούμε ας μην βάζουμε πολιτική χρειά σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Φυσικά και θα βρούμε σωστές λύσεις ε, και η ευθύνη δεν θα είναι μόνο δική σας ή μόνο δική μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ερτούκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από δική μου πλευράς. Νομίζω ότι οι προβληματισμοί είναι ανάλογοι και με τις οδικές μεταφορές. Η μεγάλη πρόκληση σε τελική ανάλυση θα είναι οι τελωνιακές δεκπαιρεώσεις και οι τεχνικές διατάξεις και πώς θα επιληθούν αν έχετε προτάσεις για το πώς μπορούν να επιληθούν όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε ευγνώμονες. Ή άλλο, θα πρέπει εμείς να κάτσουμε να σκεφτούμε λύσεις και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση για ένα συνολικό πακέτο με τον κύριο με την ε, κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και επίσης έχουμε και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ώρες, εβδομάδες και χρόνια κόπο. Έχουμε και το μεσογειακό διάδρομο, όπου εξετάζοντας κυρίως ε, τις σιδηροδρομικές ε, μεταφορές Λονδίνο, Ντόβερ, Μπέρμιγχαμ, μέχρι το, Birmingham, μέχρι το Δουβλίνο και τη Γλασκόβη. Θα ήταν κρίμα αν υπήρχαν καθυστερήσεις μέχρι το έτος 2030. Να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά σχέδια τα έχουμε αναβάλει. Θα μπορούσαμε να αναβάλουμε και άλλα. Αλλά θα πρέπει να κινηθεί και η Βρετανική κυβέρνηση αν θέλει να ωφεληθεί από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Ιδάλλως, τα πράγματα είναι και θα μείνουν δύσκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ερτούκ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τους ομιλητές, ε, διότι συχνά, όπως είπαμε, λαμβάνουμε πληροφορίες για το τι κάνετε και τα διαβάζουμε αυτά, αλλά καλό είναι αυτά να λέγονται δημόσια. Σε σχέση με αυτό που και ο Σχέρτογκ για το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά, διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, φαντάζομαι ο κύριο Χέρτο και τη επαφή με αυτού που ασχολούνται με αυτά. Είναι σημαντικό αυτό να παραμείνει στην ημέρα διάταξη, διότι είναι κρίσιμο και για τι δύο πλευρέ. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την αμοιβαία αναγνώριση ε, των ε, αδειών, τα έχουμε ζητήσει και νωρίτερα αυτό και εγώ συμφωνώ απολύτως. Ε, δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποια ένδειξη ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από την Βρετανική πλευρά. Επίσης, ε, το ίδιο ισχύει για τους κοινωνικούς κανόνες. Τώρα για το Eurotunnel. Εγώ συνήθως, ε, ε, εγώ να τον τομέα των αερομεταφορών, αλλά το Eurostar το λατρεύω και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι το Eurostar θα συνεχίσει ε, έχει από πλευράς ε, υπηρεσία στους καταναλωτές, ε, στους επιβάτες είναι ένα εξαιρετικό προϊόν γνωρίζω ε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική μεταφορά η Μάργαρη Θάτσερ η προηγούμενη Πρωθυπουργό είχε δώσει μεγάλη έμφαση, μια παλιά πρωθυπουργό μα ε, είχε δώσει έμφαση για τη και όθηση στο να δημιουργηθεί το Eurotunnel. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εμπορεύματα, ε, οπωσδήποτε πρέπει να, περνάμε, να περνάμε αυτά τα εμπορεύματα από τι οδικέ μεταφορέ και τι ε, ε μεταφορέ. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα των εμπορευμάτων. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα και όσοι θέλουν μια ε, ένα καλό αποτέλεσμα, ένα ομαλό αποτέλεσμα. Ε, το τονίζουμε αυτό όπου και όποτε μπορούμε και εσείς συνεχίστε να πιέζετε σε όλα τα επίπεδα και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα εξασφαλίσει ότι θα παρακολουθούμε στενά αυτά που συμβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Φώστερ, ο κύριος Τερλίτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και για τις παρουσιάσεις δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, από ό,τι φαίνεται καταλείπουμε κάπως ε, το θέμα της ποιότητας της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θεωρούμε ε, δεδομένο ότι η εσωτερική αγορά ε, δεν είναι εφικτή επιλογή. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν είναι. αλλά κατά κάποιο τρόπο μας, μαζί με την νέα αγορά πετάμε και τη Λονιακή Ένωση. Αλλά ίσως να πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό, διότι ε, βεβαίως ε, ε, χωρίς αυτά υπάρχουν τρόποι παρόλα αυτά να ελαχιστοποιήσουμε κάπως ε, τον αντίκτυπο, η διαφορά είναι τεράστια. Ακόμα και με την τεχνολογία, ακόμα και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, δεν θα αποφύγουμε ένα κάποιο προστατευτισμό που πάντα υπήρχε βέβαια ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να υπάρξει διάδραση δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων, των βουλευτών. Όταν έχει ξεκινήσει η συζήτηση ε, για τον Brexit πριν το δημοσίευμα, ίσως να πρέπει να έχει ακουστεί περισσότερο φωνή των επιχειρήσεων. τέλο πάντων, βεβαίω ε, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. δεν μπορώ όμω παρά να το κάνω το σχόλιο αυτό. Δεν πρέπει πάντως τώρα να εγκαταλείπουμε ε, την ποιότητα της σχέσης που θα έχουμε με τους Βρετανούς. Ε, ε, μου άρεσε πολύ η δομή σας, αναφέρομαι στην πρώτη ομιλήτρια. Επίσης, αναφερθήκατε στο θέμα των εργαζομένων, αυτών που επιχειρούν, τα στοιχεία που δώσατε είναι εντυπωσιακά. Το καθεστώς των ανθρώπων αυτών ε, είναι πολύ σημαντικό και οι δύο πλευρές γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα, αλλά ορισμένες φορές ε, καλό είναι να το λέμε, να λέμε ότι υπάρχει μια οικονομική διάσταση, μια επιχειρηματική διάσταση και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για τις βρετανικές και πολύ καλά κάνατε και το είπατε. Δεν έχω ακριβώς κάποιο ερώτημα να θέσω. Το είπα και προηγουμένως και δεν απαντήθηκε βέβαια το ερώτημα. Εσείς ε, τι αντιδράσεις προσλαμβάνετε από τους πολιτικούς εκπροσώπους ε, στην Ευρώπη αλλά και στο Λονδίνο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολιτικός ε, δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ζητήματα όπως Λωνιακή Ένωση, είτε μια ενισχυμένη είτε μια αποδυναμωμένη, γιατί δεν συζητείτε αυτό. τι αντιδράσεις βλέπετε στις επαφές που έχετε, διότι ένας έστω και μετρή, μέτρες ευθείας άνθρωπος ε, δυσκολεύεται να καταλάβει γιατί να καταλήψουμε την Λονιακή Ένωση. Ε, είναι μια βασική ανησυχία για μας ε, οι εργαζόμενοι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι και από τις πλευρές της μάχης θα πρέπει να κάτσουν και να συζητήσουν, διότι συχνά έχουμε να κάνουμε διάλογο κοφών και λυπάμαι γι' αυτό. Ευχαριστώ και ο Κράμερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρεμβάσεις και αυτό που με ανησυχεί και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερο είναι οι συζητήσει με τη, ε, μαζί σας ε, σε ό,τι αφορά και για παράδειγμα τις τρίτες χώρες, ε, την Ελβετία, την Νορβηγία. Τι γίνεται με τις συζητήσεις στον Εμένο Βασίλειο είσαστε χαρούμενοι που θα τα κάνετε όλα μόνοι σας ή μήπως ε, ε, και εσείς σκέφτεστε ότι γιατί να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, γιατί να έχουμε αυτό το κόστος. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι γίνεται στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας. Ε, μια ερώτηση. Από τι άκουσα στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία 20 χρόνια κατηγορούμε, κατηγορούσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μας εκπλήσει ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική σας οργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κράμερ και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές για να δώσουν ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. μας παρουσιάζει τα διάφορες ε, Ποιες είναι λοιπόν οι συνέπειες ε, που θα νιώσουμε στην Ευρώπη αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνείτε, γιατί είπατε ότι θα χρειαστεί μια μεταβατική κατάσταση. Πού βρισκόμαστε όμως και ποια θα είναι η αντίδραση, όπως είπε ο κ. Τελιτσικά, της πολιτικής ε, σε ό,τι αφορά τα αιτήματά σας αυτά. Γιατί προφανώς υπάρχει καταπήγον χαρακτήρας. Και το λόγο λοιπόν έχει η κυρία για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσει Να απαντήσω σε κάποια από τα ζητήματα που ετέθησαν. Καταρχάς για τους διαδρόμου ε, το TNT. Καλώς ορίζουμε κάποιες από τις επενδύσεις που έγιναν στους διαδρόμου μας και στις οδικές αρτηρίες ε, και στους συνδεδρομικούς, ε, στο συνδεδρομικό κλάδο. Και αυτό προφανώς έχει αντικτυπώ και στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Κοιτάξαμε πώς μπορούσαμε να παραμείνουμε ε, δεσμευμένοι στον ε, διάδρομο της Μεσογείου, σε ό,τι αφορά και το συνδρομικό διάδρομο και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό feedback τώρα, να σας πω ότι ήταν εξαιρετική η συμμετοχή και του Υπουργείου μεταφορών της Ευρωπαϊκής, του, του Βασιλείου και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν εξαιρετικός ο διάλογος και ήταν πολύ ανοιχτή για τις λύσεις που, προβα... που προτείναμε. Αυτό μας αναφύσε κάπως ότι λαμβάνεται υπόψη και ο τομέας των συνδρομικών μεταφορών, καθώς και μερικά συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι τροφοδοτήθηκαν στις συζητήσεις. Προφανώς έχουμε διαπραγματεύσεις υψηλού επίπεδου και θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν αυτά τα πολιτικά και μετά να δούμε τι θα γίνει, αλλά είναι θετική η εντύπωση. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στην εξέβρεση λύσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αντίδραση η πιο σωστή, η πιο ενδεδειγμένη. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η ζωή εκτός της Ελληνικής Ένωσης, κατά πόσον θα υπάρξει δυνατότητα να υπάρχει εσωτερική ελληνική διεκπαιρέωση στους, ε, στα τρένα προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα στα σύνορα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Πίπερ όσον αφορά την αναγνώριση. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα μόνο στην αναγνώριση αδειών πιστοποιητικών και αδειών ασφάλειας από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, μάλλον το αντίστροφο. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προφανώς θα αναγνωρίζουν την ε, τεχνολογία που θα υπάρχει από την άλλη πλευρά. Αλλά η βασική ανησυχία έγκυται ότι δεν πρόκειται αυτό να αρχίσει να ισχύει στην απέναντι πλευρά από την πρώτη μέρα μετά το Brexit. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα με τις άδειες ασφάλειας των επιχειρήσεων, με την άδεια των οχημάτων, με την ίδια την άδεια που φέρουν οι οδηγοί. Και έπειτα περνάμε στο δεύτερο πρόβλημα, στο δεύτερο ερώτημά σας μάλλον, αν είμαστε σε επαφή με πολιτικούς. Ναι, είμαστε σε επαφή με την ομάδα του κυρίου Μπαρνιέ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού τους λέμε, και για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο εκείνο που δεν θα έχουμε ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, ενιαίες άδειες για τους οδηγούς και το καθεξής. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει και πολύ συχνά αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε. Τώρα, όσον αφορά την ε, στάση των μελών του Μένου Βασιλείου, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας υπάρχει μια κοινή τοποθέτηση για το τι θα πρέπει να γίνει και ελπίζω πραγματικά να καταφέρουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα οποία προτείνουμε όντως να τα υλοποιήσουμε μετά τον Brexit. Ο κύριος Γκουνό. Κοιτάξτε, για το Eurotunnel δύο είναι οι βασικές ε, προτεραιότητες. Ροή των εμπορευμάτων και ασφάλεια. Όσον αφορά τη συνδρομική ασφάλεια, όπως σας είπα, έχουμε 400 με 500 τρένα καθημερινά. Ένα Eurostar έχει περίπου 900 άτομα μέσα, όσο 3-4 δηλαδή αεροπλάνα. Ξέρετε ότι ένα φορτηγό πάρα πολλών τόνων καλύπτει μια τεράστια απόσταση, μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 140 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν μέχρι το Folkestone να συνεχίσει να ισχύει και μετά το Brexit το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας. Όσον αφορά τώρα την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων και των επιβατών, έχουμε βέβαια την τεχνολογία στα σύνορα, πολλές φορές πιο σύγχρονα πλέον μέσα προκειμένου να κάνουμε ελέγχου επιβάτες. Θα πρέπει αντίστοιχα να έχουμε γρήγορα και σύγχρονα μέσα όσον αφορά τον εκτελονισμό των προϊόντων ένας τελωνιακός έλεγχος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο για ένα φορτηγό από ότι παίρνει ένα ολόκληρο κοντέινερ το οποίο φτάνει από την Κίνα σε λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε ότι ασχολούμεθα και είμαστε σε επαφή για τα ζητήματα αυτά και με τη γαλλική και με τη βρετανική πλευρά. Αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι προκειμένου να έχουμε συστήματα πληροφορικής αποτελεσματικά θα πρέπει να γνωρίσουμε ακριβώς ποιο πρόβλημα πρέπει να επιλύσουμε, ποια είναι η φύση του προβλήματος. Θα πρέπει λοιπόν εφόσον προκύψει νέος τελωνιακός κανονισμός αυτός να προκύψει το συντομότερο δυνατό και τα όσα ακούσαμε από τους προλύσαντες είναι απόλυτα λογικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς όταν καλούμεθα να δημιουργήσουμε γιγαντιαία συστήματα πληροφορικής. Συνεπώς, αναγκαστικά θα υπάρχει και μία περί, περίοδος προσαρμογής και θα πετηθεί ένας κάποιος χρόνος προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σύστημα αυτόματου εκτελονισμού και θα έλεγα ότι η σύραγγα της μάχης αποτελεί κοινοτικό και εκτιμένο. Όλοι μας φέρουμε την ευθύνη να την προστατεύσουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι στο εγγύς μέλλον που θα έχουμε και αυτοοδηγούμενα, αυτόνομα αυτο, αυτοκίνητα, τα οποία θα περνάνε από τη σύραγγα της μάχης, εμείς θα λέμε όχι, θα καθόμαστε να βάζουμε σφραγίδες στα σύνορα, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την πρόκληση αυτή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πρέπει πολύ γρήγορα να περάσουμε πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκουνό για τις διευκρινήσεις αυτές. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Πάρτ για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Προς τον κύριο Λόχμαν, καταρχάς, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την ε, διασυνοριακές ε, τεχνικές ιδιαιτερότητες τις οποίες σκεφτήξατε, υπάρχει από πλευράς ε, Βρετανικής κάποιος ομόλογος για τις συνομιλίε, για τις προετοιμασίε, ή θα ξεκινήσουν νέε διαπραγματεύσει. Ξέρω το μοντέλο το Λεβατικό και συμμετείχα σε όλη τη διαδικασία. Ήταν καινούργιε οι διαπραγματεύσει. Αυτό λοιπόν προ εσά, προ τον κύριο Γκουνό. Αναφέρατε, κύριε Γκουνό, κατά πόσον διακυβεύεται το σύστημα των τρέχων και ότι αυτό θα προκαλούσε πιο πολλά προβλήματα για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο για την ε, Μεγάλη Βρετανία. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτό επηρεάζει από πλευρά μα τι διαπραγματεύσει και του διαπραγματευτέ. Θεωρώ ότι πρόκειται για αρκετά ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε για την ποιότητα των υπηρεσιών, για τις τιμές των προϊόντων, αλλά και την όλη αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση με τους ενδεχόμενους μελλοντικούς τελωνιακούς ελέγχους. Πώς μπορούμε εμείς να καθησυχάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει σε συγκεκριμένε υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη σχέση μεταξύ Νομένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, τίθεται και ένα ζήτημα προϋπολογισμού όσον αφορά όλες αυτές ε, τις ε, διασνοριακές υπηρεσίες. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν και στα πλαίσια του προπολογισμού θα υπάρχουν στο μέλλον για το Μένο Βασίλειο συγκεκριμένε δεσμεύσει. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω πρώτα ένα σχόλιο. Ε, λόγω της μεγάλης σοφίας του Μένο Βασιλείου δεν είναι ίδιο το πρόβλημα για, τους, για τα πρόσωπα και για τα αγαθά, διότι πάντα ελέγχουν τους ανθρώπους, τα πρόσωπα, ε, οι Βρετανοί ούτως ή άλλως. Και επίσης προηγουμένως δεν αναφερθήκαμε στα λεωφορεία. Υπάρχει και η, οδική, μεταφορά, η, το, ταξίδι μέσω λεωφορείου από το Βασίλειο στην Ευρώπη. Ε, σε ό,τι αφορά τις εθνικές υπηρεσίες και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να εξετάσουμε κάπως προσεκτικά το θέμα των σιδηροδρόμων. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Επειδή είναι διαφορετική φύση οι σιδηρόδρομοι και οι οδικέ μεταφορέ και στο πώ οργανώνονται οι μεταφορέ ε, ε, και σε ό,τι αφορά του διαχειριστέ που συνήθω είναι μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί αλλά και λόγω των, των ίδιων των υποδομών, μήπω είναι πιο εύκολο να βρεθεί μία συμφωνία για τη λειτουργία μεταξύ των δύο συστημάτων του Ευρωπαϊκού και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και μήπως το Brexit θα δώσει ένα πλεονέκτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο. Αν δηλαδή το, ο σιδηρόδρομος ε, θα, θα, θα αποκτήσει πλεονέκτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα για το Eurotunnel, ε, ερώτημα προς τον πρόεδρο Γκουνό, το Brexit απειλεί το νομικό καθεστώς, το διεθνές αυτό νομικό καθεστώς της υποδομής του Eurotunnel. Ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ. Ο Βέρνερ Κούν. Καλημέρα Βέρνερ. Η εσωτερική αγορά και η Τελεμιακή Ένωση προφανώς ε, πάνε μαζί και στον ε, σύγχρονο κόσμο τα χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε την ενιαία μας αγορά. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρέ καλά θα κάνουν να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Ήταν πάρα πολύ αβαντκάρτη το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων με το τέταρτο πακέτο. Πάντα υπήρχε διάκριση του δικτύου και τη ε, διαχείριση. Ε, Έπαιζε μεγάλο ρόλο αυτό. Όντω λοιπόν πήγαν τα πράγματα έτσι και θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τις διαπραγματεύσει. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Και κοιτώντα, ε, το είπε και προηγουμένω ο συνάδελφο Κράμερ, τι συστήματα αποτελούν το πρότυπο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία είναι όντω η Νορβηγία θα κάνουμε τα ίδια με την Ελβετία σε ό,τι αφορά τους σιδηροδρόμους. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι είναι καθαρός φορές, με 5,6 δισεκατομμύρια το χρόνο το μεγάλο φαινόμενο βασίλειο. Αλλά σε ό,τι αφορά όχι του κύκλου εργασιών, αλλά την καθαρά την εκτακεφαλή εισφορά ανακάτοικο είναι 89 ευρώ το χρόνο, ενώ στην Ορβηγία είναι 78, χωρί να έχουν καν επίτροπο, χωρί να αναμειγνύονται στι Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Να σκεφτούμε λοιπόν και αυτή την διάσταση σε ό,τι αφορά τη μελλοντική διαμόρφωση. Σα ευχαριστώ πολύ, η κυρία Άντερσεν. Ναι, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την δημόσια υπηρεσία, είναι καλό να εξετάσουν το θέμα αυτό των μεταφορών οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό δεν γίνεται απαραίτητα σε πολιτικό επίπεδο. Τι, σκοπό σου έχετε λοιπόν έτσι ώστε το, το θέμα να είναι πιο ψηλά, έτσι ώστε οι πολιτικοί θύνοντε να δώσουν σημασία στο θέμα των μεταφορών. Πολύ καλό ότι έχουμε εδώ ένα εκπρόσωπο τη Eurotunnel. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Φώστερ από αυτού. Η Μάγκρα θα πρέπει να πω ότι προτιμούσε έναν οδικό, ένα οδικό τούνελ, έτσι όχι ένα σιδηροδρομικό. Μια και εδώ, ε, όμως, τι γίνεται με τις ε, ε, υπηρεσίες της Deutsche Bahn. Είναι πολύ καλό βέβαια ότι υπάρχει το κύριο Στάρα, αλλά θα πρέπει να μπορεί και η Deutsche Bahn να περνάει τρένα από το, το τούνελ. Ε, για όσου είναι αντίθετοι στον ευρωσκεπτικισμό, είναι περίεργο που πλέον λέγεστε Get Link και όχι Eurotunnel. Μπορείτε να μας πείτε ότι εξακολουθείτε να είστε ε, φιλοευρωπαίοι, όπως πάντα beaucoup, Madame Anderson. Monsieur c'est à vous. Ο Κι Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για την παρουσίαση πολύ χρήσιμη. Το ερώτημά μου αφορά την Eurotunnel. Ε, βεβαίως η Τελωνιακή Ένωση αφορά μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρεται. Ε, αυτό θα έχει λοιπόν επιπτώσεις ε, και για τις μεταφορές ε, αγαθών και αυτό πρέπει να είναι ανησυχητικό, μεταφορές εμπορευμάτων. Ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όμως και σε ό,τι αφορά το, τη μεταφορά επιβατών. Ευχαριστώ τον κύριο Τέιλορ. Ο Βιμ Βαντενκάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Πρώτη. Προ την κυρία Ράιτ μου αποστήλατε μία επιστολή στις 13 Νοεμβρίου του 2017, στην οποία και αναφέρεται ότι 41.000, υπήκοοι από τις 27 χώρες μέλη εργάζονται στους συνδρομού της Μεγάλης Βρετανίας. Πρακτικά, πώς το φαντάζεστε τι πρακτικά προβλήματα παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά τις άδειες παραμονής, άδειες εργασίες, διαβατήρια. Τι θα πρέπει να προβλέψουμε. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Λόχμαν για την περίοδο μετάβασης. Ρώτησα και στον τομέα των οδικών μεταφορών πώς πρόκειται να οργανωθούμε. Εσείς τι προτιμάτε, να συνεχίσουν να υφιστάνονται οι τρέχοντες κανόνες μέχρι ότι υπάρχει οριστικό Brexit για το οποίο εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή να υπάρχουν κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις, το οποίο προφανώς θα περιπλέξει τα πράγματα πολύ. Θέλετε να το τοποθετηθείτε. Και τέλος, προ... στον CEO της Eurotunnel. Υπάρχει κίνδυνος ε, η συνοριοφυλακή φυλακή και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα προκειμένου να μπλοκαριστεί η ελεύθερη μεταφορά και διακίνηση. Ελπίζω να μην δίνω ιδέες στους Βρετανούς, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε και ρεαλιστές. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις διάφορες απόψεις και ερωτήσεις που εκφράσατε. οι 41.000 Ευρωπαίοι υπήκοοι που εργάζονται στους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας, τι συνέπειες θα υποστούν. Μιλάμε για δικαιώματα των πολιτών. Και το θέμα της μεταβατικής περίοδου. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί αν υπάρξει μεταβατική περίοδος, γιατί αν δεν υπάρξει μεταβατική περίοδος, η συζήτηση αλλάζει. για τον κύριο Κούνο. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του Brexit. Θα αλλάξει το καθεστώς, το δικό σας. Και ποια είναι τα συστήματα τα οποία φαντάζεστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το Brexit. Γιατί αν όπως ε, διατείνεται η Τρέζα στην Αγγλία, η Αγγλία βγει από, τον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ενιαία Αγορά και από την Τελεανική Ένωση, τι θα γίνει. Τι θα σημαίνει αυτό για σας. Αν θα θέλετε να απαντήσετε σε τρία λεπτά, παρακαλώ. Έχετε και πιο πολύ ώρα από ό,τι προηγουμένως. Ευχαριστώ. Σε έξι σημεία νομίζω ότι θα έπρεπε να απαντήσω γρήγορα. Πρώτον, θέλουμε να παραμείνουμε εταίρος της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Θεωρούμε ότι η Βρετανία μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ σε διάφορες διαδικασίες, διακανονισμούς και διευθετήσεις. Το είχαμε κάνει αυτό και στο παρελθόν. Ξέρω ότι κάποιοι θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε υψηλό βαθμό επίπεδο, όσον αφορά δηλαδή το ζήτημα της μελλοντική μας συμμετοχής στον οργανισμό αυτό. Θα θέλαμε πάντως να συνεχίσουμε να αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του οργανισμού αυτού. Τώρα για τους 41.000 υπηκόους ε, των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται στους Βρετανικούς σιδηροδρόμους, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένας πολύ καλός εργοδότης. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους, πιο ταλαντούχους, 20.000 είναι τα προγράμματα κατάρτισης και θέλουμε να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό, θέλουμε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τους πιο προκισμένους εργαζόμενους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η τελική συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται και διαμένουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ να σας δώσω λοιπόν μια συγκεκριμένη απάντηση. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα για τη μετώπιση όλων των εργαζομένων, όχι μόνο των πιο ειδικευμένων εκπαιδευμένων και το πιο ταλαντούχων που εργάζονται στο σιδηροδρομικό τομέα, αλλά και αυτούς που έχουν άλλες δεξιότητες, γλωσσικές και άλλες. Νομίζω ότι θα πρέπει και αυτοί να, έχουν, να χαίρουν ενός ε, ξεκάθαρου απλού συστήματος απασχόλησης. Ξέρετε ότι ε, οι ε, Βρετανικοί σιδηροδρόμοι έχουν θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά πρωτοπόροι, και αυτό το διαβάζουμε και στο τέταρτο σιδεροδρομικό πακέτο, θέλουμε να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό και να συνεχίσουμε να έχουμε τα ύψιστα αυτά επίπεδα ικανοποίηση των πελατών. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι σε ορισμένες από τις αρχές του τέταρτου πακέτου του σιδεροδρομικού και δεν θα θέλαμε λόγω του Brexit να υπάρξει αλλαγή σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τώρα τους Δημοσίου υπαλλήλου. Ε, εξαιρετική ήταν η στάση του. θα ήθελα να του ευχαριστήσω, αλλά να απόκειται τελικά στου πολιτικού ε, να λάβουν τι τελικέ αποφάσει. Συνεργαστήκαμε με υπουργού από τα αρμόδια υπουργεία, θέσαμε τα ζητήματα αυτά σε τακτική βάση είμαστε σε επαφή μαζί τους, ε, επομένως ε, βλέπετε ότι ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους σε όλα τα επίπεδα, κρατώντας τους σιδηροδρόμους ψηλά στην ατζέντα. Επίσης είμαστε σε επαφή με εκπροσώπους και από άλλους τρόπους ε, μεταφορών και όπως ακούσαμε φάνηκε και από το πρώτο πάνελ έχουμε κοινέ ανησυχίες και με τον τομέα των οδικών αλλά και των θαλασσίων και των αέριων μεταφορών. Μία τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω όσον αφορά το ζήτημα των επενδύσεων στους σιδηροδρόμους. Όντως ε, είχαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους Βρετανικούς σιδηροδρόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πολλές επενδύσεις και σε εγχώριο επίπεδο. Επενδύσεις που πηγαίνουν στις υποδομές πάνω από 50 δισεκατομμύρια τα επόμενα 10 χρόνια θα επενδυθούν στην υποδομή των Βρετανικών σιδηροδρόμων. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να προωθείτε, να συνεχίσει να προωθείτε να προωθούνται οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ, να βνοούνται σε σχέση με άλλου τρόπου μεταφορών. Αυτό είδαμε στο παρελθόν, αυτό θέλαμε να δούμε και στο μέλλον. Ο κύριο Μπλόκμαν τώρα έχει το λόγο, θα είμαι σύντομο να απαντήσω σε κάποιε ερωτήσει όσον αφορά το ζήτημα τη αναγνώριση και τις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις ρυθμιστικές αρχές του Μένου Βασιλείου. Αυτό θα θέλαμε να κάνει η RDG με το Eurostar καθώς επίσης και με άλλους παράγοντες από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου. Να καταφέρουμε να έχουμε μία αυτόματη ενιαία αναγνώριση μεταξύ των αδειών που υφίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των αδειών των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαντώ έτσι και στο ερώτημα του κυρίου Ρικέ. Ναι, θα πρέπει να είχαμε μια συμφωνία στην αυτή που υπάρχει για τις οδικές μεταφορές που να καλύπτει όλες τις μορφές ε, μεταφορών και στον τομέα των σιδηροδρόμων, έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση Brexit. Και να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Βάντεν Κάμπ. Για μα η μεταβατική περίοδο είναι σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη φυστάμενο καθεστώ σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο όπω έχει σήμερα για ένα όσο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά το Brexit. Αυτό το δανεικό Και μπορεί έπειτα να πάρει μια άλλη μορφή που θα μπορούσαμε να τη βαφτίσουμε ακόμα και συμφωνία για χερσαίες μεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα μας ρωτήσατε ποια θα είναι το μέλλον των τελωνίων σε σχέση με τις νέες αυτές διαδικασίε, Μα ήδη από τώρα πρέπει να μετασχηματίσουμε λίγο τις διαδικασίε που ακολουθούμε, διότι Ξέρετε ότι θα πρέπει ε, να, να περάσουμε από τις γραπτές ε, έντυπες διασαφήσεις στις ηλεκτρονικές τελεινικές διασαφήσεις. Έχουμε το NCTS, ένα νέο μορφότυπο ηλεκτρονικό που ακολουθούμε στα τελωνία. Πολλές λοιπόν οι προκλήσεις ήδη από τώρα όσον αφορά την προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος και βέβαια αυτό ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τώρα οι τελεινιακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται και στα σύνορα στο μέλλον, α γίνονται εκεί, αλλά α μην επινοήσουμε πάλι ένα νέο σύστημα, α συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε το NCTS και σε χερσαία σύνορα εφόσον αυτά προκύψουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκουνό τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όντως, το Ενωμένο Βασίλειο δεν ήταν ποτέ στο χώρο Σέγγεν, άρα γινόντουσαν πάρα πολλοί έλεγχοι και για τα λεωφορεία, πάρα πολλά από αυτά περνάνε από τη σύραγγα της μάχης και ξέρετε ότι γίνεται ήδη ένας πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός έλεγχος, πολύ καλύτερος από ό,τι στα αεροπλάνα. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο των σιδηροδρόμων, κοιτάξτε, το μέλλον είναι η διαλειτουργικότητα. Αν πραγματικά θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη σύραγγα τη μάχη και να περνάνε από αυτήν και γερμανικά τρένα τη Deutsche Bahn, ε, θα πρέπει προφανώς να διατηρήσουμε το όραμα της διαλειτουργικότητας όπως το έχουμε σήμερα και να φτάσει βέβαια αυτό το όραμα αυτό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ότι την Άνοιξη του 18 θα έχουμε μια διασύνδεση πλέον Λονδίνο-Άμστερνταμ είναι ήδη ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τη γεωγραφική εν μη τι άλλο παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τώρα την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Πάλι μέσω της σύραγγα της μάχης έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη θετική αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας και να σας δώσω εδώ πέρα δύο παραδείγματα. Όλα τα οχήματα τα οποία κατασκευάζονται στο Μένο Βασίλειο ουσιαστικά απαρτίζονται από εξαρτήματα επιμέρους τα οποία έχουν κατασκευαστεί στη Γερμανία και τα οποία περνάνε επί από τη σύραγγα της μάχης και συναρμολογούνται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα άλλο αντίστροφο τώρα παράδειγμα. Ο Σολομός από την Σκοτία που μας αρέσει σε όλους. Ένα 95% του Σολομού αυτού περνάει από το τούνελ αυτό, φτάνει στην Μπουλόνιου Σιωμέρα και εκεί πέρα συσκευάζεται, τη χάνει περαιτέρω μεταποίησης και στη συνέχεια επιστρέφει και για πόλη... στο Ηνωμένο Βασίλειο περνώντας πάλι από το τούνελ. Ξέρετε ότι έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τα πιο αποτελεσματικά οικονομικά συστήματα για να αποκριθούμε στις ανάγκες των καταναλωτών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε, τα θετικά αποτελέσματα δηλαδή που έχουμε πετύχει. Τώρα, κάποιες πιο γενικές παρατηρήσεις. Η τρομοκρατία, προφανώς ζήτημα επώδυνο, αναφέρθηκε αυτό από κάποιου. αποτελεί ε, πολύ σημαντική ανησυχία και μέλημα του Eurotunnel. Συνεργαζόμαστε εδώ πέρα με διάφορους αρμοδίους από διάφορες χώρες. Οι ειδικοί μας λένε ότι τη στιγμή που επινοήθηκε και δημιουργήθηκε το ε, τούνελ αυτό, είχαμε την περίοδο τότε της δραστηριότητας του IRA IRA ε, σχεδόν κάθε εβδομάδα εκρήξει του Ηνωμένο Βασίλειο, άρα είχαν ληφθεί υπόψη, αν θέλετε, όλες αυτές οι ανησυχίες τρομοκρατία που υφίστανται ήδη από τότε και προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να διευκολύνουμε και τη μετακίνηση των σιδηροδρόμων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαρωτές, σκάνερς στην είσοδο και στην, στην είσοδο μάλλον της σύραγγας της μάχης προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη σάρωση και ένα πιο ενδελεχή έλεγχο των άμαξοστοιχειών. Τώρα όσον αφορά το όνομα της επιχείρησής μου Ξέρετε ότι η επιχείρηση Eurotunnel είναι η επιχείρηση που μέχρι στιγμή διαχειρίζεται τη σύραγγα της μάχης. Κατά 95% βρισκόμαστε στην Ευρώπη, δεν πρόκειται να καταλήψουμε λοιπόν την Ευρώπη. Αλλά ξέρετε ότι είναι η μητρική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ένα 75% των επενδυτών στην μητρική εταιρεία είναι ξένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άνθρωποι από τις ΗΠΑ, η Κίνα, διάφορες ασιατικές χώρες, η Αυστραλία και μου κάνει εντύπωση που στην Αυστραλία καταφέρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι επενδυτέ τουλάχιστον εκεί πέρα, να καταλάβουν καλύτερα τα όσα διακυβεύονται αυτή τη στιγμή για το Eurotunnel από ό,τι το καταλαβαίνουμε εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την μητρική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθότι όπως σας είπα η μητρική εταιρεία είναι αυτή που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Αποφασίσαμε για το λόγο αυτό λοιπόν να περάσουμε από το όνομα Eurotunnel στο όνομα GetLink. Και έχει δημιουργηθεί και μια ανεργειακή πλέον διασύνδεση που φέρει το όνομα ELEC Link και θέλουμε μέσω του ονόματος GetLink να συνεχίσουμε να συνδέουμε το Νομένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να καταχειροκροτήσουμε τους καλεσμένους μας. Πραγματικά η παρεμβάση σας ήταν ε, υψή τη ποιότητος και ειλικρινά σας ευχαριστώ που μας διαθέσατε τόσο χρόνο και επαναλαμβάνω ότι θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Μεταφορών διότι ε, εμείς ε, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ε, τομιακή ανάλυση πλέον του Brexit και θα θέλαμε να είχαμε τη συμμετοχή σας και στο μέλλον. Τώρα, συνοψίζοντας πολύ σύντομα, θα ήθελα να σας πω ότι θίξαμε διάφορα ζητήματα σήμερα το πρωί συζητώντας τον Brexit και τον αντίκτυπο που θα έχει στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, είδαμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο αίσθημα ανησυχίας και αβεβαιότητας. Το θίξατε αυτό πάρα πολύ. Έχουμε δύο χερσαία σύνορα, την Ιρλανδία, αλλά χερσαίο σύνορα αποτελεί τελικά και σύραγγα της μάχης. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει με τους τελωνιακούς δασμούς, με την επιπλέον γραφειοκρατία, με όλους αυτούς διακανονισμούς που θα πρέπει να ισχύουν στο μέλλον. Όλα αυτά θα πρέπει να τα θέσουμε πραγματικά στο κέντρο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αποφανθούμε οριστικά για όλα αυτά τα ζητήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη τουλάχιστον φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί αυτό ο πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι μεταφορέ στο μέλλον μετά το Brexit. Συνεχίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα στι 3 η ώρα το μεσημέρι όπου θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα ζητήματα της μερίσιας διάταξης. Καλή όρεξη σε όλους. Καλό μεσημέρι.